Παρακαλώ τοποθετήστε όλοι τις κάρτες. Right. Are we having an anonymous vote, or is that meant to be green? Right. The, the, the vote is open, so as soon as you've. Λοιπόν, αρχίζει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Βάλτε τις κάρτες και ψηφίστε.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 like Right, at the moment we've got 38 members who have got their cards plugged in and we've only got 28 who've pressed a button. Μόνο 28 έχουν πατήσει το κουμπί και σας παρακαλώ εάν πραγματικά θέλετε να περάσουμε στις πραγματικές ψηφοφορίες βάλτε τις κάρτες για να κάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Και έχει και υπερβολικό θόρυβο στις άλλες.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 We now have 40 cards. Λοιπόν, 40 έχουν βάλει τις κάρτες τους και 32 έχουν ψηφίσει. Όσοι έχουν τοποθετήσει τις κάρτες, παρακαλώ να ψηφίσουν για να ελέγξουμε. Okay, can I just, for, the, for those that might be confused, I'm hoping you επαναλαμβάνω, ελπίζω να έχετε τοποθετήσει τις κάρτες, να έχετε ψηφίσει ώστε να ελέγξουμε ότι το μηχάνημα του καθενός δουλεύει. 41 έχουν τοποθετήσει τις κάρτες, στους 34. Μα είναι αναμένο το μικρόφωνο μου. Ας προσπαθήσω με ένα άλλο μικρόφωνο. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Α, ωραία. Right, can you hear on that one? Oh, great. <laughs> Τώρα που βάλαμε την τουντούκα ακούτε καλύτερα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, 44 έχετε τοποθετήστε. Κάντε σε 34 μόνο πιέσατε και το κουμπί. Οπότε παρακαλώ τους 10 που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία να πατήσουν και το κουμπί. Σαράντα Τέσσερις, δύο ακόμη. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος δεν το έχει κάνει, αλλά δεν πειράζει. Καλά είμαστε και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε για τις διαφανείς δεξαμενές έκθεση Swinburne. Συμβιβαστική H πρώτα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I, λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 80 καταπίπτει περνάμε στη συμβαστική και η λατινικό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική L υπέρ. Η K ψηφίστηκε. L υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική N, όπως Νίκος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική O, αντιβρό ναι, υπέρ. Α, βέβαια, είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία αυτή. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Δεν έχω καταλάβει τι ψηφίζουμε, λέει ο ε. πρόεδρος. Α, μάλιστα. Πρώτο τμήμα της O, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 123. 123 υπέρ κατά αποχές, νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική π υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 140 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα την 140. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Βλέπετε το αποτέλεσμα. 21 ψήφι υπέρ, 24 κατά. Τροπολογία 141 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε και αυτό. 141. Ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα και επειδή νομίζω δεν είπα ότι λίγη ψηφοφορία, καλό θα ήταν να ξανά ελέγξουμε την 141. Τώρα από το ΕΛΚΑ έχουν ψηφίσει πιο πολύ από όσους έπρεπε. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ που ψηφίζει. Τώρα είμαστε εντάξει, ψήφισαν όλοι, άρα τώρα εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τώρα, τροπολογία 142, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 143, υπέρ. Κατά. Αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστικές υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε εφόσον το ζητάτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 29 κατά. Τροπολογία 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω θα την θέσω σε έλεγχο. 166. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 152 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική U Α, ναι, έχετε δίκιο. Το, πρέπει να ψηφίσουμε το πρωτότυπο, το αρχικό κείμενο του 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάλι πηγαίνουμε στην 164 τροπολογία. Ή όχι. Μα εγκρίθηκε η U. Εντάξει. Λοιπόν, έχει εγκριθεί η συμβαστική υγιού και πηγαίνουμε στην τροπολογία 164. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160... Ποιο είναι το πρόβλημα? Εγκρίθηκε. Το είπα. Τροπολογία 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παράγραφη 22 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Εντάξει, θα το ελέγξουμε. Το αρχικό κείμενο λοιπόν της παραγράφη 22. Λοιπόν, αφού είχε ζητηθεί έλεγχος θα το ελέγξουμε. Εγώ είχα δίκιο. Εγκρίθηκε. Συμβαστική Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται θα το ελέγξουμε όμως το δεύτερο τμήμα Έχετε ψηφίσει όλοι. Εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στη συμβιβαστική W. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 175, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 κατά πίπτη. Τροπολογία 177 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 183 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Y. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. Με προφορική τροπολογία που προσθέτει τις λέξεις where appropriate. Για να καλυφθεί η εταιρική κατάσταση, αν κάποιος ε, έχει αμφιβολίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 191 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε. Κάνω ένα πρόβλημα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Το πρώτο τμήμα μπορεί να προσθεθεί σε συμβιβαστική Β. Είναι συμβατά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα. Εκεί, για την 30 θα έλεγα τώρα. I don't know what anybody is contesting. Δεν ξέρω που διαφωνείτε, ποιος διαφωνεί. Τέλος πάντων, εγώ πηγαίνω στην τροπολογία 30 τώρα. Η πρόεδρος ε, έχει δίκιο, μου αρέσει αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που έχω δίκιο. Λοιπόν, τροπολογία 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική η e, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, γιατί λέει εδώ ότι καταπίπτει 42, τέλος πάντων. Πηγαίνω συμβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, α, συγγνώμη, πρώτο τμήμα της F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής F, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αλλά ας το ελέγξουμε, γιατί υπήρξε κάποια σύγχυση. Α, εντάξει, εγκρίνεται. Απλά κάποια περίεργα, έτσι, κάποιες περίεργες χειρονομίες Τροπολογία 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 43 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. We are now on agenda item 14. Πάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ? Κάζα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, εκθέση Κάζα. Υπέρ της τροπολογίας 2. Κατά. Ωραία. Ξέρετε που είμαστε. Είμαστε στην έκθεση Κάζα, τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Έχουμε προφορική τροπολογία στην 4 από τους πράσινους. Αντικαθιστούμε το φόρο με το φραγμούς του στη φορολογία. Όχι, δεν υπάρχει προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε την 4 όπως είχε στην αρχική της μορφή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ναι, συνεχίστε να ψηφίζετε. Ωραία. Εγκρίνεται. 44 με 2 κατά και για το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ψήφισατε όλοι. 40 υπέρ, 2 κατά. Ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Κάσα. Πάμε στο σημείο 15 της ημερησίας τώρα. Ψηφοφορία για την γνωμοδότηση ΣΥΡΠΑ Πιετικάινεν. Κυρία Πιετικάινεν, θέλετε να λάβετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 9. Προφορική, η προφορική συγγνώμη τροπολογία του ΕΛΚ στο δεύτερο τμήμα, δηλαδή της ε, χωριστής ψηφοφορίας, εάν είναι κατάλληλο, δηλαδή ή όπου είναι κατάλληλο το if appropriate, και που μιλάμε δηλαδή για την κατάλληλη νομοθεσία κλπ. κλπ. Αυτό ήθελα μόνο να σας πω σε σχέση με αυτή την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Ναι, θα το κοιτάξουμε όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Είσαστε πάντως έτοιμοι. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, ήταν το αρχικό κείμενο. 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται νομίζω και αυτό λέει πρόεδρος. Θα το ελέξω αν θέλετε. Άρχεται η ψηφορία. Πέραση ψηφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο, παράγραφος 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 9, στο τρίτο τμήμα, όταν φτάσουμε, ξεκινάμε με το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία. Στο τρίτο τμήμα τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Να προσθέσουμε τις λέξεις, τις λέξεις if appropriate. Συμφωνείτε με αυτή την προφορική τροπολογία, το if appropriate. Αν είναι κατάλληλο, αν κρίνεται κατάλληλο όπου χρειάζεται, ποιε είναι υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε, λέει ο Πρόεδρος. Has everybody Right. Ωραία. Περαστή πληροφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ της 10 ξαναλέω. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1 σημείο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Συμβασμός Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 καλύπτεται, οπότε περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφορία για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι, 35 υπέρ, 5 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Πιτικάινεν. Okay, Συνάδελφοι, θα πρέπει να αποφασίσουμε πριν πάμε στην ψηφορία. Όπως θα μάθατε από email, είχαμε ένα αίτημα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης να περιλάβουμε το σχέδιο γνωμοδότησής τους εδώ και το οποίο δεν είχαν ευκαιρία να ψήφισουν ακόμα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Γι' αυτό μου ζητήθηκε να εξετάσω κατά πόσο θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε εδώ. Θέλω λοιπόν τη σύμφωνη σας γνώμη για να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση επειδή αυτή ακόμα δεν έχει ψηφιστεί στην Επιτροπή τους. Οπότε διαδικαστικά θα πρέπει να σας ρωτήσω κατά πόσο επιθυμείτε να ψηφίσουμε για θέματα που αφορούν την, ε, την ομοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης υπό τον όρο βεβαίως ότι θα προληφθούν μόνο όσα είναι συμβατά με τη δική μας νομοδότηση. Αν έχετε αντίρρηση δεν θα ψηφίσουμε. Αλλά είπα στον πρόεδρο, στο Προεδρείο της Επιτροπής Απασχόλησης ότι θα το θέσω στην Επιτροπή μας για να αποφασίσει η δική μας Επιτροπή. Πού πήγατε? Ποιος ζήτησε το λόγο? Είμαι έτοιμη να ακούσω τον εισηγητή και ο μηχανισμός που θα ακολουθούσαμε θα ήταν προφορικέ τροπολογίε, οπότε υπάρχει λύση. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου παρακαλώ και για αυτό το θέμα τρεις σύντομε παρατηρήσεις, παρότι γνωρίζω ότι δεν είναι ασυνήθιστο πριν από την ψηφοφορία να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να επισέλθω στα θέματα ουσία. Το μόνο που θέλω είναι σύντομα να επιχειρηματολογήσω και να πω πώς τον πίνακα ψηφοφορίας, πώς κατέληξα στις συστάσεις του καταλόγου ψηφοφορίας από πλευράς μου. Διότι πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι, όχι τόσο εδώ στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στις συναρμόδιες επιτροπές, ε, έχουν κάποιες ε, αυταπάτες για αυτά τα θέματα και πρέπει να πω κάποιε κάποιες παρατηρήσεις γι' αυτό. Επί της ουσίας ε, είχαμε ψηφοφορία σήμερα το πρωί και έχουμε τροπολογίες επ' αυτών που λόγω αρχής θα πω όχι και θα απορρίψω επειδή πολύ πιεστικά ήταν ε, τα περιθώρια τα χρονικά. Δεν είχα καμιά ευκαιρία να δω την ουσία του θέματος. Και επειδή θέλω στο τέλος να έχουμε μια συναφή συνεκτική γνωμοδότηση ως κοινοβούλιο, δεν μπορώ να δεχθώ τέτοιες προτάσεις. Κάποιοι από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου είπαν να προτείνεις κάτι το οποίο πάει πολύ πιο μακριά. Τότε θα έχουμε μια καλύτερη βάση διαπραγμάτευσης ως κοινοβούλιο. Συνάδελφοι, δεν έχουμε καθόλου κακή θέση διαπραγμάτευσης ή καλή θέση διαπραγμάτευσης. Δεν έχουμε καμία θέση διαπραγμάτευσης και πρέπει να το γνωρίζουμε. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε, εντάξει δεν παζαρεύουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι κατά το μάλλον ή να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και τίποτα άλλο. Γιατί είναι μόνο διαβούλευση και είναι και κάτι λιγότερο από διαβούλευση κιόλα για παράδειγμα, στην εξωτερική υπηρεσία, διπλωματική υπηρεσία, είχαμε την δυνατότητα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας τις θέσεις μας έναντι του Συμβουλίου να τις περάσουμε, όπου είχαμε μόνο διαβούλευση. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μια νομική βάση σύμφωνα με την οποία δεν διαβουλευόμαστε εμείς. Είπε το Συμβούλιο εθελοντικά θέλουμε ως Συμβούλιο να έχουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου και έτσι στην πρώτη, ψήφιση, πρώτη ψηφοφορία θα ψηφίσουμε για να αλλάξει αυτή η νομική βάση. Αλλά και πάλι αυτό είναι στο χέρι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο μπορεί να πει δεν υπάρχει γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, δεν μας ενδιαφέρει το θέμα περαιτέρω. Με άλλα λόγια πρέπει, αν θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα πράγματα κάπως, πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ως Ευρωκοινοβούλιο. Και γι' αυτό θέλω να σας πω το εξής. Αυτά τα οποία πρότεινα εγώ, ήδη για την ημερομηνία κιόλα, είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ μας. Επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε ακόμα πιο πέρα και μου είναι συμπαθής αυτή η προσπάθεια που θέλουν να κάνουν. Αλλά σε αυτούς τους συναδέφους ε, μπορώ να αναφέρω κάποιους άλλους στην αίθουσα που για την ημερομηνία του 2018 και πέρα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν έχει να ένα νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα εντυπωσιαστούν αν έχουμε μια σαφή πλειοψηφία υπέρ της σύστασής μας. Γι' αυτό η σύσταση ήταν 2018 παρότι θα προτιμούσα να είχαμε μια άλλη λύση και μια άλλη ημερομηνία. Η δεύτερη παρατήρηση ένα τέτοιο κανονισμό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων δεν πρέπει να τον θεωρούμε ως ευχολόγιο, ως ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο οποίο κρέμονται πολλά δώρα που δεν έχουν καμιά θέση εδώ. Έχουμε από την Περιφερειακή Επιτροπή πολλέ τροπολογίε. Πρέπει να επιχειρηματολογήσω και να πω γιατί θέλω να τι καταψηφίσω. Συμπαθητικό είναι το αίτημα και σε σχέση με τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ μετά το 2013-2014 να ενισχυθούν αυτέ οι περιφέρειε. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση αυτό με τον κανονισμό για επιδοτήσει και ενισχύσει ω θέμα. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Μια τρίτη παρατήρηση. Αν έχουμε τώρα θέμα σύγκρουσης με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Είμαι ο πρώτος που είμαι υπέρ μιας τέτοιας σύγκρουσης, αλλά να γνωρίζουμε δεν έχουμε δυνατότητα να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Το σημείο είναι το εξής. Κάνουμε, συντάσσουμε μια γνωμοδότηση. Το Συμβούλιο μπορεί να πει δεν μα ενδιαφέρει καθόλου η γνωμοδότησή σας. Μόλις πιο πριν το είχα αναφέρει. Το Συμβούλιο πρέπει με ειδική πλειοψηφία να αποφασίσει γι' αυτό. Αν το κάνει αυτό και το δεχτεί, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πει ναι εντάξει αποσύρουμε τη δική μας πρόταση, θα υποβληθεί μια νέα πρόταση από εμά. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε πρέπει ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβούλιο. Αλλά τότε δεν θα αλλάξει καθόλου η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι, να το γνωρίζουμε. Να δώσουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να τροποποιήσει κάτι, να αλλάξει κάτι, όπου δεν θα απολέσει το κύρος της και θα τηρηθούν τα προσχήματα. Ε, διότι μπορούμε να πούμε, μπορεί, μπορεί να αναφερθεί παραμένουμε σε αυτή την πρόταση και δεν αλλάζουμε τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα αλλά θα πρέπει αν πούν ότι εντάξει για την ημερομηνία 2014 τη δεχόμαστε δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι όμω ε, πρέπει να δουν πώ θα κινηθούν, πώ θα ελιχθούν και γι' αυτό είχα πει ότι στον πίνακα ψηφοφορίας είχα διατυπώσει συστάσει για να αποστείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα καλύτερο θα ήταν να διαπραγματευόμαστε, αλλά δεν έχουμε διαπραγματευτική θέση. Αυτό δεν γίνεται και έτσι πρέπει να ψηφίσουμε αυτά. Αυτό όμω δεν είναι το πρόβλημα μα. Ε, έχετε αντίρρηση. Ωραία. Ο αντιπρόεδρο έχει αντίρρηση. Άννα Νομίζω ότι έτσι θέτουμε ένα προηγούμενο να εξετάσουμε γνωμοδοτήσεις Οπότε θα θέλαμε να θέσουμε ένα προηγούμενο εδώ. Ωραία. Ωραία. Είπα προηγουμένω ότι ο μόνο μηχανισμό που θα ακολουθούσαμε θα ήταν οι προφορικέ τροπολογίε. Οπότε τέρμα έχει λήξει το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κύριο Λάγκεν. Ζητώ τον λόγο για την ομάδα του ΕΛΚ. Θα ήθελα σε σχέση με τον εισηγητή και την αντιπρόεδρο να δώσω δίκιο και να πω δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία για μη αποφασιστέντα σχέδια. Εξάλλου κατά τα άλλα στις τροπολογίες της ΕΚΟΝ έχουμε όλες τις εναλλακτικές πιθανές λύσεις που σκιαγραφούμε και στις ψηφοφορίες σήμερα το πρωί που είχα συμμετάσχει στην Επιτροπή Ήτρε ήταν τέτοια η καθυστέρηση που δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη αυτές οι τροπολογίες. Και εδώ δεν πρόκειται για θέμα συναπόφασή μα, αλλά για μια γνωμοδότηση έναντι κανονισμού του Συμβουλίου. Και πρέπει έγκαιρα να λειτουργούν τα πράγματα και να λειτουργήσουν. Δεν έχει νόημα να αναβάλουμε τα πράγματα, δεν θα ασκήσουμε τότε καμιά επιρροή. Γι' αυτό παρακαλώ με τον κατάλογο τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας στην Επιτροπή Ήτρε έχουν συμπεριληφθεί αλλά δεν είναι πλήρη διότι μόνο το μεσημέρι δόθηκαν τα κείμενα. Τίθεται ένα αποφασιστική σημασία θέμα εδώ και πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Ο εισηγητής έχει αν μπορώ να το διακηρύξω έτσι, μια προφορική τροποποίηση, ένα προφορικό αίτημα για την ημερομηνία 2018. Εντάξει, εμείς, εγώ ο ίδιος, είχα τροπολογία για το 2020 και άλλοι εξίσου και αρκετοί συνάδελφοι κιόλας. Το ερώτημα τώρα είναι, αν εμείς θα δεχτούμε και θα επιτρέψουμε η τροπολογία του συναδέλφου Ράπκαη 2018 να είναι η ημερομηνία ως η πιο μακριά, η πιο απόμακρη και έτσι να ψηφιστεί πρώτη αυτή. Τότε θα είχαμε σαφή πλειοψηφία γι' αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα εμείς η ομάδα μας, η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα είναι υπέρ του 2018 ως πρότασης και να επιχειρηματολογήσω, να το εξηγήσω γιατί. Ο Αλμούνια, ο κύριος Αλμούνια, μετά από σε βάθος επιστημονική και νομική εξέταση, πρότεινε το 2018 ως ημερομηνία. Και γι' αυτό το, η Επιτροπή, για την Επιτροπή το 2018 την έχουμε στο πλευρό μας ως εταίρο με αυτή την πρόταση του 2018 παρότι με, οποιοδήποτε άλλο, με, οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Αν γίνει δεκτό αυτό και αυτό θα έλεγα να γίνει 2018 να είναι η ημερομηνία θα ήμουν πρόθυμος στις δικές μου τροπολογίες για το 2020 να τις αποσύρω. I think uh, I, see people being happy with... Βλέπω ότι συμφωνείτε, μάλλον θέλετε να προχωρήσετε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Λάγκη. Θα το αντιμετωπίσουμε όταν φτάσει η ώρα. Περάμε τότε στην ψηφοφορία. Πρώτα η προφορική τροπολογία του εισηγητή στο 1. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 67 ήτρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 ήτρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 69 ήτρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε τώρα, στην τροπολογία 55 υπέρ, 57 συγγνώμη υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έτσι νομίζω. Όχι, να το ελέγξουμε. Απλά είδα να σκόνται πολλά χέρια. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε τελικά. Η 58. Είναι ταυτόσιμη με την 59. Α, όχι. Πηγαίνουμε στην 59. Α, είναι αυτή που έχει αποσυρθεί, μάλιστα. Άρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε τώρα. 14 ήτρε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 ήτρε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ. 63 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 63. Τροπολογία 62 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται και αυτή αλλά θα το ελέγξουμε. Μισό λεπτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται αυτή. Μάλλον όλοι ψηφίζετε στην κόψη του ξηραφιού. Λοιπόν, όλες οι άλλες καταπίπτουν. Μα το είδατε το αποτέλεσμα. Όχι. Μα ήταν 22 υπέρ, 21 κατά. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Υπήρχαν δύο παρόντες βουλευτές που δεν ψήφισαν. εγώ το είπα, να πατάτε τα κουμπιά γρήγορα. Αν εσείς δεν συγκεντρώνεστε και δεν με ακούτε, ε, είναι θέμα των ομάδων. Δεν είναι δικό μου. Right, we're now going on to... 87, 87 ήτρε τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 ρέτζι, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 65, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν κάποιες και πάμε στην τροπολογία 69. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 ήτρε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 ρέγγι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι υπόλοιπες μέχρι μέχρι τη 18 Ήτρε. 18 Ήτρε λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73 αποσύρθηκε. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τρεις από εσά δεν έχουν ψηφίσει. Ένας ψήφισε. Λοιπόν, 28 κατά, 16 υπέρ. Κάποια στιγμή ότι αντιπρόεδρο θα με πιστέψει, τέλος πάντων rejected. It was rejected, yes. It was clearly, you said 28 against 11 or something like that. It was clearly rejected. Then we go to 11. Then we go to 11. I don't know what your problem is. No, there is no problem. No, it says 19 falls. If adopted, rest except IPTRI 19 falls. Λοιπόν, μετά από αυτή την μικρή συνεννόηση γιατί τα έχω λίγο χάσει. Πάμε στην τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία να ελέγξουμε την 11. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Ένας, ε, τώρα έχει ψηφίσει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία. Ένας από το ΕΛΚ να αποσυρθεί. Εγκρίνεται λοιπόν η 11. Τώρα τροπολογία η 11 εγκρίνεται. Έτσι και τώρα πηγαίνουμε στην 19. 19 Ήτρε. Δεν υπάρχει αυτή η τροπολογία. Okay, we are now going to vote on... Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την τροπολογία 28. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι ο κατάλογο ψηφοφορία ε, καταρτίστηκε κάπω απότομα, ε, τελευταία στιγμή και είναι λίγο περίεργη, τέλο πάντων. Λοιπόν, τροπο 28. Περ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 21 ήτρε υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 105 ήτρε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 ρέτζι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε την 78 γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο. Άλλοι δύο. Ένας. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. 81 τροπολογία υπέρ. 81 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε Λάγκεν, ε, σας παρακαλώ να καθοδηγήσετε. Οδηγήστε, καθοδηγήστε τα μέλη της ομάδας σας. We, Ήτρε 108 τροπολογία. Ήτρε 108. Τι λέτε. In Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 αποσύρθηκε Ρέτζι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε οι υπόλοιπε καταπίπτουν μέχρι την 19 τροπολογία 19 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 αποσύρθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αυτή 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ήτρε συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήτρε 33 υπέρ κατά απόχέ απορρίφθηκε ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ρέτζι 4 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίφθηκε Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ρέτζι 7 ε, υπέρ Ρέτζι 7 7 Ρέτζι υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Άλλοι τρεις για να ψηφίσουν και να ολοκληρωθεί. Η τελευταία ευκαιρία και κλείνει η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η ισοψηφία 19-19 απορρίφθηκε. Πάει αυτή. Αιτιολογική σκέψη 3. Προφορική τροποποίηση από πλευρά εισηγητού είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Όλα τα άλλα καταπίπτουν. Μέχρι την 26. 26 λοιπόν. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 27 αποσύρθηκε ή 44 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ρέτζι 10 υπέρ μια στιγμή κατέπεσε αυτή όχι Ρέτζι 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Αποσύρθηκε αυτή. Ωραία. Τροπολογία 46 τώρα. Υπέρ. 46. Ήτρε 46 παρακαλώ. Πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, Ήτρε 46 είπαμε. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ρέτζι 13 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ρέτζι 13. Αυτή ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Δύο ακόμα που μπορούν να ψηφίσουν. Τελευταία ευκαιρία πριν λήξει η ψηφοφορία. 28 εναντίον 17 υπέρ. Κατα... Απορρίφθηκε. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 34 τώρα, ναι η 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πηδάμε τώρα σε κάποιο άλλο σημείο. 38 τροπολογία. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ρέτζι 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την Ρέτζι 16 άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ Ένας παραπάνω συμμετείχε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ για το ότι αποσυρθήκατε. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Ρέτζι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά ελέγχουμε. Όχι. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Εισηγήτου υπέρ. 4. Σελίδα 22 εκεί βρίσκομαι. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 Ρέτζι υπέρ κατά μια στιγμή καταπίπτει επειδή η προηγούμενη είχε την κιανή εγγραφή καταχώρηση καταπίπτει λοιπόν η 43 μπορούμε να την ψηφίσουμε τη 43 43 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τοπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 48 με προφορική τροποποίηση που δεν την έχω εδώ Δεν χρειάζεται όμως αυτή πια. Γιατί είχαμε μια άλλη προφορική τροποποίηση στο σκεπτικό 3, στην αιτιολογική σκέψη 3 και δεν χρειάζεται εδώ να επαναλαμβάνεται η προφορική τροποποίηση. Και να ψηφίσουμε έτσι όπως ε, είχε προταθεί από τον συνάδελφο. Να υπερψηφίσουμε λοιπόν αυτή τη θέση. Ψηφίζουμε λοιπόν την, την αρχική τροπολογία, χωρίς την προφορική τροποποίηση. Εντάξει, αρχική τροπολογία 48, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Ρέτζι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήτρε 65 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήτρε 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το τελικό κείμενο που ψηφίζουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε 32 υπέρ. 8 εναντίον, 5 αποχές. Επίσης, παρότι δεν έχουμε αυτό στον κατάλογο, πρέπει να ψηφίσουμε το ψήφισμα ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν και πάλι ψηφοφορία για το ψήφισμα. Για το ψήφισμα, εντάξει. This is a vote on the Ψηφίζουμε το ψήφισμα με αυτή την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξέρω ότι δεν το έχετε στα έγγραφά σας αλλά μια και άλλαξε, τροποποιήθηκε το κείμενο. Δύο ακόμα να ψηφίσουν ένας και λίγη ψηφοφορία. Τελική ευκαιρία κλείνει η ψηφοφορία. 32 υπέρ 8 εναντίον, 4 αποχές ε, εγκρίθηκε. Uh, Κύριε Ράπκα, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ απλά μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για άλλη μια φορά να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα γιατί εδώ τώρα έχουμε δύο ή τρεις ε, ας το πω έτσι πιο ασύμβατες θέσεις μη συναφή. Αυτό εξηγείται επειδή την τελευταία στιγμή είχαμε τόσες πολλές τροπολογίες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε, από την Επιτροπή Ήτρε. Υπάρχουν τρεις ασυμβατότητες. Πρέπει μέχρι την Ολομέλεια να χτενίσουμε το κείμενο για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ήθελα να το αναφέρω αυτό για τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει αυτό. We've got three more items on the agenda, so don't go. Έχουμε ακόμα τρία θέματα στην ημερήσια, μην φύγετε. Δύο λεπτά διάλειμμα για να βρούμε πού βρισκόμαστε. Okay, everybody, if we could resume seats. Right, we have, we have three items on the agenda. Έχουμε ακόμα τρία σημεία στην ημερήσια όπου θα έχουμε ελπίζω τους εισηγητές short selling και credit default swaps και μετά καθηγητή πιστός εξαγωγών και κατευθυντήρες γραμμές ή και αξιολόγηση. Θέμα αυτό το τελευταίο που το αναβάλαμε από το πρωί. Θα στραφώ λοιπόν προς τους ηγητές για το short selling και τα credit default shops. Αυτοί που συζητάνε παρακαλώ να συζητήσουν έξω γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα τη δουλειά μα. Όσοι θέλουν κουβεντούλα να βγουν έξω παρακαλώ. Thank you. Is it quiet enough yet? Thank you, Pascal. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Έχω την τύχη και την χαρά να είμαι εισηγητή τη του Κοινοβουλίου. Να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν για το γεγονό ότι δεν είχα χρόνο να σας μοιράσω ένα γραπτό έγγραφο με τις θέσεις που θα σας παρουσιάσω τώρα. Το χρονοδιάγραμμα που επιλέξαμε είναι έτσι πολύ στενό. Καταρχήν επειδή έχουμε να κάνουμε ένα κανονισμό οπότε πρέπει να εγκριθεί σύντομα και στη συζήτηση με τους διάφορους κοιόδης θα θέλαμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που συμπίπτει με αυτό του Συμβουλίου ώστε να έχουμε ανταλλαγές ευφυείς και καρποφόρες όσο γίνεται. Αυτά λοιπόν για το λόγο για τον οποίο δεν είχα το χρόνο σας δώσω ένα πρώτο έγγραφο. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Θα έχετε την έκθεση που θα συντάξω γύρω στις 22-23 του Νοέμβρη, στις επόμενες 15 μέρες δηλαδή. Μια επενθύμηση για το πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν που ανάγεται στα μέσα του Σεπτέμβρη. Είχαμε δύο φάσεις πολιτικών αντιδράσεων και των ρυθμιστών όσον αφορά το social selling. Πρώτα, το 2008 μετά την πτώση της Lehman Brothers, διάφορες ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών αγορών έλαβαν αποφάσεις για την απαγόρευση του short selling για διάφορες μετοχές και μετά μια δεύτερη φάση, ένα δεύτερο κύμα για τα credit for swaps τα κρατικά. Την άνοιξη του 2010 θα θυμάστε είχαμε το θέμα του ελληνικού χρέους και είχαμε διάφορες ε, πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αντιδράσεις από τις ρυθμιστικές αρχές που αποφάσισαν και πάλι να απαγορεύσουν το short selling. Ε, στη Γερμανία ιδιαίτερα πώς θα θυμάστε. 2008 λοιπόν και άνοιξη 2010 αυτά που έγιναν μας έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ώστε τα μέτρα που λαμβάνει μια χώρα να ακολουθούνται και από άλλες χώρες ώστε να μην υπάρχει μια αποσπασματική και κατακαιρματισμένη ενιαία αγορά που δεν θα λειτουργεί. Δεύτερο συμπέρασμα που μπορούμε να συνάξουμε από αυτή την εμπειρία είναι ότι κατά διάρκεια αυτών των δύο περίοδων χρειαστήκαν περισσότερη διαφάνεια. Επειδή θυμάστε το, την άγγιση του 2010 χρειάστηκαν διάφορες εβδομάδε τους ε, Ευρωπαίους για να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβαινε με, τα, με το εθνικό χρέος κάποιων χωρών μελών. Όλοι λοιπόν κατέληξαν στο ότι χρειάζομαστε ένα κοινό καθεστώς πιο διαφανές ώστε να παρακολουθούμε με τρόπο πιο ακριβή τους κινδύνους. Και αυτό οδήγησε βεβαίω την Κομισιόν στις 15 του Σεπτέμβρη να καταθέσει ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο καλύπτει διάφορα θέματα. Δεν θα τα αναφέρω τώρα όλα σε αυτή την ταχεία παρουσίαση με τρία σημεία κλειδί. Πρώτο σημείο κλειδί η διαφάνεια, μετά το marking και μετά το όριο κοινοποίησης, κοινοποίησης δηλαδή στις ρυθμιστικές αρχές και προς το σύνολο των παραγόντων της αγοράς. Δεύτερος πυλώνας του κειμένου της Κομισιόν, η βούληση για να πλησιώσουμε καλύτερα το naked ναι short selling, τις γυμνές ανοιχτές πωλήσει, όπως λέμε, υποχρεώνοντας τους ε, φορείς να εντοπίσουν τους τίτλους που θα ε, πολλούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα παράδοσης στη συνέχεια ώστε πραγματικά να υποχρεώνονται να δανειστούν τον τίτλο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να πουλήσουν. Μετά έχουμε και το θέμα της διάρθρωσης μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Για αυτά τα τρία λοιπόν σημεία κλειδί, ως εισηγητής, θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση, δίνει κάποιες απαντήσεις τις οποίες θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσες, και ως εισηγητής θα προσθέσω δύο θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται ή δεν ε, αντιμετωπίζονται άμεσα από την Κομισιόν, δηλαδή κατά πόσο πηγαίνουμε μέχρι την απαγόρευση του naked short selling, απαγόρευση εφενός και πρόταση της Κομισιόν αφετέρου, που δεν είναι ακριβώς απαγόρευση, και μετά για το θέμα των CDS, των ακάλυπτων, uncovered CDS δηλαδή, όπου η Κομισιόν δεν προτείνει την απαγόρευσή τους και θα επιχειρηματολογήσω όπως έκανα με τους σκιώδεις λέγοντας για ποιο λόγο, για ποιους λόγους ότι η απογόρευση των uncovered CDS μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση. Πρώτος πυλώνας λοιπόν διαφάνεια. Η γενική προσέγγιση της Κομισιόν βρίσκεται σύμφωνο. Υπάρχουν δύο ε, διατάξεις, μάλλον δύο συστήματα τα οποία είναι συμπληρωματικά. Το marking που αφορά το γενικό σύστημα των ε, ροών ώστε να διασφαλίσουμε στους ε, ε, ρυθμιστές πλήρη γνώση του τι θα πρέπει να καλύπτουν όλων δηλαδή των συναλλαγών, κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο και θα επιτρέψει στους ρυθμιστές να ξέρουν τι γίνεται. Επιπλέον έχουμε ένα σύστημα κοινοποίηση και αυτό το σύστημα κοινοποίηση είναι βέβαιως χρήσιμο αλλά έχει και αυτό τα ωριά του, δηλαδή αφενό ε, πρόκειται για ένα σύστημα κοινοποίηση το οποίο γίνεται ημερησίω, οπότε έχουμε πληροφορίες δηλαδή ε, μια φορά την ημέρα τα μεσάνυχτα ε, για τον υπόλοιπο χρόνο δεν ξέρουμε τι γίνεται, γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε το marketing και ένα άλλο στοιχείο τη κοινοποίηση είναι τα όρια και αν η συμμετοχή της αγοράς είναι λίγο πιο κάτω από τα όρια ακριβώ για να μην υπάρχει κοινοποίηση τότε ο ρυθμιστή δεν έχει καμία πληροφορία στη διάθεσή του σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει κανεί όταν κάνει παρεμβάσει στην αγορά επειδή ακριβώ βρίσκεται λίγο κάτω από το όριο που χρειάζεται κοινοποίηση. Οπότε καταλάβαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε αυτέ τι δύο διαδικασίε που προτείνει και προβλέπει η Κομισιόν. Διάφορα επιχειρήματα ακούστηκαν από τότε σε σχέση με αυτές τις προτάσεις, ιδιαίτερα για το marking και το επιχείρημα που ακούμε περισσότερο είναι το κόστος. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό βεβαίω και αυτό ακριβώς στην πρότασή μου λέω δεν γίνεται να επιβάλλουμε το marking στο σύνολο των αγορών ας πούμε τρεις μήνες μετά ας πούμε την εφαρμογή του κανονισμού. Αντίθετα μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πρόταση για το marking και θα μπορούσαμε να την ενσωματώσουμε στην ενημέρωση του συνόλου των συστημάτων και των υποδομών πληροφόρησης ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς το κόστος του μάρκετινγκ να γνωρίζουμε ακριβώ δηλαδή το κόστο του μάρκετ και να λέμε στι διάφορε αγορέ: Κοιτάξτε, έχετε ένα, δύο, τρία χρόνια και θα συζητήσουμε πότε τέλο πάντων για να σωματώσετε, για να υιοθετήσετε αυτό το σύστημα στι υποδομέ τη αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και η απαραίτητη υποδομή πληροφορική ώστε να γνωρίζουμε ακριβώ βέβαια το κόστο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι το CDS Corporate Δηλαδή μίλησα προηγουμένως για την διαφάνεια. Η διαφάνεια αφορά βεβαίως τις ε, μετοχές και τα σεντές στα κρατικά. Όμως θα ήμασταν υπέρ, υπό το όνορο βέβαια ότι αυτό δεν θα ήταν βαρύ για τους ε, παράγοντες. Θα ήμασταν υπέρ λοιπόν του γεγονότο οι ρυθμιστές να έχουν στοιχεία και για το corporate CDS επειδή οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην αγορά ε, με σκοπό τη χειραγώγηση αφορούν κυρίως τα SEDAs, τα, τα κρατικά, αλλά και τα corporate. Τώρα, τι γίνεται με την πραγματική οικονομία, ε, τι διακυβεύεται εκεί. Αν έχουμε ενδεχόμενες χειραγωγήσεις για τα corporate CDS, τότε θα έχουμε αύξηση της τιμής των CDS. Η αύξηση της τιμής των CDS θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων του χρέους των επιχειρήσεων, δηλαδή των, της με την οποία χρηματοδοτούνται και βεβαίως η επένδυση σε αυτή την περίπτωση θα κοστίσει περισσότερο στις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι καλό για την δραστηριότητά τους επιχειρηματική και την απασχόληση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε κατ' νου ακριβώς τι γίνεται και στην αγορά των corporate CDS ώστε να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους που περιέγραψα. Δεύτερος πυλώνας είναι το θέμα της απαγόρευσης ή όχι του naked short selling και naked CDS. Προσωπική μου θέση είναι να πούμε ότι το short selling αυτό καθε αυτό δεν θέτει προβλήματα. Αντίθετα, το net naked short selling είναι αυτό το οποίο είναι πιο κερδοσκοπικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν συμβάλλει σχεδόν καθόλου στην πραγματική οικονομία ούτε και στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές ενώ αντίθετα έχει πολλούς κινδύνους και η σχέση τιμή κίνδυνος οι πλεονεκτήματα κίνδυνος, αν δούμε το naked short selling, μου φαίνεται ότι είναι μάλλον υπέρ της απαγόρευσης του naked short selling, επειδή το πλεονέκτημα αυτής της ε, τεχνικής δεν είναι και τόσο μεγάλο, δηλαδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε τελείως τις ε, δραστηριότητες αγοράς, αλλά λέμε ότι παίρνουμε τα καθαρά και οροσκοπικά στοιχεία και προσπαθούμε να τα περιορίσουμε. Ένα άλλο στοιχείο είναι πλαισίωση. Υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν που αφορά τις κυρώσεις που προτείνονται σήμερα. Δεν υπάρχει ένα αρμονισμένο σύστημα κυρώσεων ε, στην Ευρώπη, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τις προτάσεις της Κομισιόν όπως αναφέρονται, δηλαδή με κυρώσεις οικονομικές και να υπάρχει και υποχρέωση ε, αγοράς των τίτλων, bailing out procedure. Το ξαναλέω, αυτά είναι οι δύο πυλώνε του συστήματο με τι κυρώσει που προτείνει η Κομισιόν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, έστω και αν δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε ό,τι κάνουν και αυτέ, ε, το κάνουν από το 2008, μειώνοντα σημαντικά τα προβλήματα που αφορούν την ε, έκδοση των τίτλων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε εδώ αυτό το παράδειγμα. Τώρα για τα κρατικά CDS και τα uncovered CDS, τα γυμνά που λέμε στα γαλλικά δηλαδή, naked, η Κομισιόν δεν προτείνει να τα, ακυρώσουμε, να τα απαγορεύσουμε για τους ίδιους λόγους που λέγαμε για τα corporate. Γιατί το κάνουμε αυτό. Οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης. Τα CDS αποτελούν έναν τρόπο, δηλαδή αν εσείς αυξήσετε την τιμή του CDS, αυτό οδηγεί απαραίτητα στην αύξηση του κόστους του επιτοκίου, δηλαδή την αύξηση του κόστους του δανεισμού για την ολόγω χώρα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επιτρέψουμε σε έναν οικονομικό παραγότο, ο οποίος δεν κατέχει τίτλο σε μια χώρα να αγοράσει ένα CDS ε, για το δανεισμό μιας χώρας οπότε σε αυτή την περίπτωση είτε ε, δέχεστε, αποδέχεστε τον κίνδυνο και έχετε τον τίτλο είτε δεν έχετε αυτό τον τίτλο οπότε δεν έχετε τίποτα το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί και το οποίο σχετίζεται άμεσα με το κίνδυνο πτωχεύση της χώρας τότε δεν έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε το CDS Κάποιοι θα απαντήσουν βεβαίω ότι αυτό επιτρέπει να καλύψουμε ένα κίνδυνο που δεν αφορά μόνο τι χώρε, αλλά αφορά και τι επιχειρήσει μια χώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν επ' αυτού και άλλα οικονομικά εργαλεία ή χρηματοοικονομικά εργαλεία. Εξάλλου, έχουμε ακούσει εδώ στην πολλά για την χρηματοοικονομική καινοτομία. Τα οποία όμω, εργαλεία, τα οποία όμως δεν διέρχονται απαραίτητα από την αγορά CDS, επειδή των κρατικών CDS, επειδή τα CDS τα κρατικά έχουν αυτή τη ιδιαιτερότητα όταν τα αγοράζετε τι κάνουν, αυξάνουν την τιμή του CDS, οι αγορέ των CDS, οπότε το κόστος αντιμετωπίζει ένα ψηλότερο κόστος δανεισμού. Πρόκειται λοιπόν για ένα εργαλείο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό στόχο της κάλυψης δηλαδή του κινδύνου μια χώρα, επειδή το δεχόμενο πτώχευση δεν αποτελεί κίνδυνο για τον αγοραστή, του CDS και υπάρχουν και άλλοι παράγοντε ε, στην αγορά και οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πολλά άλλα εργαλεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα ζητούσα ως εισηγητή την ε, απαγόρευση των ε, naked CDS. Τώρα, νομίζω ότι το σημείο ισορροπία στην πρόταση της Κομισιόν μεταξύ των Εθνικών Αρχών και της ΕΣΜΑ μου φαίνεται θετικό Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν επιθυμούσε το Κοινοβούλιο και υπάρχει η δυνατότητα για την ΕΣΜΑ να έχει την τελευταία λέξη ώστε να εναρμονιστούν τα συστήματα λήψη αποφάσεων τα εθνικά. Βρισκόμαστε δηλαδή εδώ σε μια λογική πραγματικής ευρωπαϊκής εναρμόνισης. Αντίθετα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα για μια χώρα μέλος να κάνει περισσότερα από αυτά που θα προτείνει ο τελικός κανονισμός. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε ένα είδος ε, περιθωρίου επικουρικότητας το οποίο θα είναι και πιο φιλόδοξο, πιο ευέλικτο από τον κανονισμό. Οπότε νομίζω ότι το τελευταίο σημείο ισορροπίας που παρουσιάζει η Κομισιόν εδώ μου φαίνεται σωστό, είναι αποδεκτό και θα το υποστηρίξω. Βλέπω ότι και στο Συμβούλιο κάποιες χώρες μέλη θέλουν να εξασθενήσουν, να κάνουν πιο αδύναμα τα σημεία κλειδιά αυτής της πρότασης κανονισμού και εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε την ευθύνη να αντισταθούμε τουλάχιστον πριν ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που επίσημα θα ξεκινήσουν τον ε, Δεκέμβρη ενδεχομένω και Γενάρη-Φλεβάρη. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε ε, τις απόψεις μου, συνάντησα και τους διάφορους κοιόδης και ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρα συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στρέφομαι στους κοιόδης τώρα. Πρώτα του ΕΛΚΑ. Μάκος, εσύ. vielen Dank, Το πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο εισήγητη, διότι πράγματι έγκαιρα ήρθε σε επαφή και στους κοιόδης εισήγητες ε, ζήτησε να συζητήσουμε τα θέματα. Το χαιρετίζω αυτό, αυτή τη μορφή συνεργασίας. Ολοκληρώνοντας ένα θέμα, μια εργασία. Μια εκπρεμή παρατήρηση θέλω να κάνω. Από όλες τις συζητήσεις που είχα για αυτό το θέμα, τίθεται αυτό ως ερώτημα. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε. Δημιουργήθηκε κάτι στην αγορά και σίγουρα υπάρχουν που σίγουρα εμπεριέχονται κάποια ενδιαφέροντα προϊόντα. Τέλος, όμως ποιος χρειάζεται στο τέλος τέλος αυτά τα προϊόντα. Τα χρειαζόμαστε. Διαφορετικές απαντήσεις μπορούν να δοθούν ανάλογα με το τι είναι short selling σε σχέση με μια συναλλαγή. Κάποιος πουλάει κάτι το οποίο δεν είναι ιδιοκτησία του και διαθέτει κάτι το οποίο δεν έχει στην ιδιοκτησία ενός άλλου. Θέλουμε αυτά να τα ρυθμίσουμε και μέσα σε ένα πλαίσιο να λειτουργούν. Τίθεται το ενδιαφέρον ερώτημα λοιπόν. Τι γίνεται εδώ και πρέπει να απασχοληθούμε με αυτό. Σαν κάποιος που είχε την τιμή να γεννηθεί στο Augsburg όπως ο Μπέτορ Μπρέχτ, είναι καλύτερο να ιδρύσει κανείς μια τράπεζα, θέτω το ερώτημα, ή να ληστέψει κανείς μια τράπεζα. Ερώτημα. Αυτό σε σχέση με το τι θα μπορούσε να είναι έγκλημα <laughs> έχει ενδιαφέρον Γι' αυτό αυτό το θέμα θα πρέπει να το προσεγγίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση κάπως. Ο εισηγητής θέτει κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα και εγώ δεν έχω κάποια καθοριστική τελεσίδικη άποψη. Αν δούμε όμως ε, τι γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το marking, τι έχει υπόψη της. Αν κάποιος ζητάει marking και δεν έχει τίποτα υπόψη του με αυτό, και είπε ο εισηγητής ότι θα μπορούσε να φανταστεί ότι για μια χρονική περίοδο θα μπορούσε να εισαχθεί κάτι τέτοιο για να τηρηθούν οι δαπάνες σε κάποια όρια. Αν όμως εισαχθεί κάτι τέτοιο, ποιος θα έχει όφελος στο τέλος τέλος από αυτό ή ποια πρόσθετη αξία θα απορρέει από κάποιες πληροφορίες που θα έχουμε για κάποιους μέσω της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή που ούτως ή άλλως ε, στο εμπορικό δελτίο αναφέρονται. Τίθεται το ερώτημα, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες νέου και όλα αυτά συνδέονται με το θέμα των αξιών κατοφλίων. Αν κάνουμε κάτι σε ένα σημείο, θα πρέπει και σε άλλο σημείο να δώσουμε συνέχεια. Ή διαφορετικά όχι, για να είμαστε συνεπείς. Αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται νομίζω, δεν συνάδουν. Από τη μία πλευρά κάνει εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται στις κανονικές ε, ομαλές συναλλαγές, από την άλλη πλευρά όμως κάνει κάτι που δεν χρειάζεται κανείς και δεν χρειάζεται. Marking, δηλαδή ο προκαθορισμός ε, αυτών των ε, ε, συναλλαγών. Πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο ή όχι. Δεν έχω τελεσίδικη προκαθορισμένη άποψη, αλλά πρέπει να τα δούμε. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και πρέπει να αντιπαρατεθούμε με αυτό. Αν θέλουμε να συμφωνήσουμε να εισαχθεί μια τέτοια, ένας τέτοιος καθορισμός, ε, τότε θέλουμε, πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει με τις πληροφορίες. Το να έχουμε μόνο πληροφορίες και να ξέρουμε κάτι, αυτό επαρκεί. Πιστεύω πως δεν επαρκεί και ότι οι δαπάνες είναι υπερβολικές για κάτι τέτοιο και δεν δικαιολογούνται. Και θέλω να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μεταξύ μας. Μετά το θέμα των κατοφλίων τιμών. Πού βρίσκονται οι σωστές τιμές κατόφλια. Μέχρι στιγμής κανένας δεν έδωσε πιστικά στοιχεία, αριθμητικά πιστικά στοιχεία και για τη συζήτηση και την προκατακτική εργασία του Σεζάρ, αν τα δει κανείς όλα αυτά, πάλι δεν έχουμε κάποιες πιστικές πληροφορίες. Δηλαδή ψάχνουμε για βελόνα στάχυρα, το πω έτσι. Τι γίνεται για να συναγάγουμε ένα συμπέρασμα. Και το νόημα του εγχειρήματο πρέπει να είναι στο τέλος τέλος να μεριμνήσουμε μέσω υψηλών τιμών κατοφλίων όλα να παραμένουν κάτω από αυτές τις υψηλές ε, τιμές κατοφλίου ή να έχουμε τέτοιες δαπάνες που θα προκαλούνται λόγω χαμηλών τιμών κατοφλίων που δεν θα δικαιολογούν πλέον την προσπάθεια. Δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί να υπάρξει marking καθορισμός, προκαθορισμός και μετά από πέντε χρόνια να δούμε αν άξιζε τον κόπο ή όχι και μάλλον και με βάση αυτή, την ε, ρύθμιση να δούμε ότι δεν πήγε κάτι καλά. Θα πρέπει λοιπόν λογικά να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να ενταθούν, αν είναι αναγκαία ή όχι. Ο εισηγητής δεν έχει επίσης θίξει ένα άλλο θέμα, το οποίο το θεωρώ αξιόλογο. Τι γίνεται δηλαδή με τους απασχολούμενους, με τις συναλλαγές εκείνες που γίνονται σε μία μέρα ε, αυθημερών και που σε σχέση με την έννοια της μη καλυπτόμενης ε, συναλλαγής ε, δεν ανταποκρίνονται αλλά μέσα σε μια μέρα καλύπτονται για μια συγκεκριμένη μέρα. Αυτό τι γίνεται σε σχέση με μια χώρα όπου αυτά μπορούν με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν και σε άλλη ίσως όχι. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Για το CDS, τα Credit Default Swaps, μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Να υπάρξει μια διασφάλιση, μια ασφάλεια έναντι, ας το πω έτσι, πτώχευσης ή κατάρρευσης ομολόγων. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις προτάσεις. Για οποιονδήποτε έχει ασχοληθεί με κρατικά ομόλογα γνωρίζει περί πρόκειται και να μην υπάρχει κάποια κερδοσκοπία όταν κάποια κρατικά ομόλογα δεν εξυπηρετούνται πλέον ή όταν οδηγούμαστε σε μια κατάρρευση και μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά και να δούμε σε σχέση όχι μόνο με αυτόν τον κανονισμό αλλά και σε ένα πιο σφαιρικό πλαίσιο. Έχουμε τη Συμφωνία Βασιλείας 3 και τι γίνεται σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Αν κατάλαβα σωστά τα πράγματα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη για την ε, αποκατάσταση κεφαλαίου από πλευρά τραπεζών σε περίπτωση ζημιάς που θα έχει προκληθεί ε, και στο τέλος τέλος και στην τελευταία σύνοδο από αυτήν απορρέει το ποιες πιθανές αλλαγές συνθήκης θα πρέπει να συζητηθούν και πάλι εδώ είχαμε την τιμή να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, ε, τον κύριο Γιουνκέρ. Και πάλι τίθεται εδώ και ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Τι θα γίνει με τον ρόλο για παράδειγμα της εποπτικής αρχής σε σχέση με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Έχει νόημα, ιδιαίτερα όταν θέλουμε κάποιες απαγορεύσεις να επιβάλλονται. Μέσα σε μια ενιαία αγορά, πώς μπορεί κάτι τέτοιο να λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις και τα δύο φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν και οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Εδώ παρότι ίσω δεν ανταποκρίνεται από την, στην προέλευσή μου που είμαι Γερμανός είμαι της κεντρικής ε, διαχείρισης ε, και όχι υπέρ της ομοσπονδιακής ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό αν θα μπορεί να είναι εφικτό πρέπει να το συζητήσουμε τι είναι το καλύτερο και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης θα είναι θέμα ποια θα είναι τα ποσοστά και ποιες αρμοδιότητες θα έχουν οι εθνικές ε, αρχές εποπτείας και τι θα γίνεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή. Πρέπει και αυτά να τα ξαναδούμε αν θέλουμε να πορευθούμε μια τέτοια πορεία. Χρειαζόμα, θα χρειαζόμαστε από πλευρά ΕΣΜΑ περισσότερες εξουσίες ή ε, διαφορετικά λιγότερες, ε, λιγότερες εξουσίες στην ΕΣΜΑ και περισσότερες από πλευρά των εθνικών αρχών σε ένα ομοσπονδιοποιημένο θα έλεγα πρότυπο Γι' αυτό είμαι ευγνώμων για το ότι ο εισηγητή έχει υποβάλει ένα χρονοδιάγραμμα που πραγματικά είναι αποτελεσματικό γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει κίνδυνο ε, το Συμβούλιο να μα ξεπεράσει σε σχέση με την κοινή μα θέση. Δεν θέλουμε με κανένα τρόπο, πώς να το πω έτσι, να μας επιβληθεί κάτι. Ναι, αγαπητέ Ρόμπερτ, είσαι αισιόδοξο εσύ και δεν μπορώ να κατανοήσω ότι κατέληξε στου σοσιαλιστέ όντα αισιόδοξο, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι μια άλλη ιστορία αλλού το είχαμε αυτό και ότι ξαφνικά το Συμβούλιο ε, επαρκέστηκε με μια κοινή θέση όπου το κοινοβούλιο δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί και δεν ήταν αποτελεσματικό. Γι' αυτό πρέπει πολύ έγκαιρα, πρόημα, όπως προτείνεται και από τον εισηγητή να δράσουμε και να μπορέσουμε μέχρι τέλους να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει με αυτή μας τη θέση και να κάνουμε διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα. Το Κοινοβούλιο σε αυτά τα σημαντικά θέματα ως πεδίο πρέπει να μπορέσει να υιοθετήσει μια σαφή θέση. Εμείς ως ΕΡΚ θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τηρηθεί το δεσμευτικό αυτό χρονοδιάγραμμα, το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, ώστε έγκαιρα να έχουμε καθορίσει μια θέση ως Κοινοβούλιο και με αυτή να τεθούμε αντιμέτωποι με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Ρομπέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πασκάλ Καμφέν για τον τρόπο με τον οποίο φέρει σε πέρα σε αυτή την κοινή δουλειά. Αφού τον άκουσα μπορώ να πω ότι είμαι σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο μήκο κύματο ε, με τον εισηγητή. Ο Μάρκος Φέρμπερ έθεσε κάποια πολύ ε, σημαντικά ερωτήματα. Και το πρώτο μάλιστα ζήτημα που έθεσε ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Χρειάζεται πραγματική οικονομία, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία συζητούμε. Είπε ο Μάρκος ότι πρέπει να προσπαθήσουμε τάχιστα να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μην ε, βρεθούμε προεκπλήξεις με μια κοινή θέση του Συμβουλίου. Δεν είναι, θεωρώ ότι υπάρχει ε, τέτοιος κίνδυνος ε, και πραγματικά θα με εξέπλησε ιδιαιτέρως αν ε, στις αρχές του επόμενου έτους είχε ήδη καταλήξει σε κοινή θέση το Συμβούλιο με βάση αυτά που ακούω από τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Μάλλον το αντίθετο θα συμβεί ως συνήθως. Για ποιο λόγο, γιατί για μια ακόμη φορά συζητάμε για κάτι που έχουμε και πάρα πολλά να κερδίσουμε και πάρα πολλά να χάσουμε. Τι μας έδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση, ότι όλα αυτά τα ωραία εργαλεία και οι τεχνικές πωλήσεων ιδίως αν υπάρξουν εντάσεις στην αγορά, μπορούν να οδηγήσουν σε πτωχεύσεις ή ιονή πτωχεύσεις. Και αυτό έχει τεκμηριωθεί πολύ καλά και σε μια έκθεση του Κογκρέσου του Αμερικανικού για την Μπίριστον, στη Λέμαν Brothers που τελικά πτώχευσε στην ΑΕΓΕ που έγινε κατά ε, την τελευταία στιγμή η επιχείρηση διάσωσης ε. στην έκθεση, στη μελέτη επιπτώσεων η Κομισιόν αναφέρει ότι δεν είναι διαφανής η αγορά αυτό των παραγόγων και θα το χαρακτήριζα εφημισμό αυτό. Η Κομισιόν, όπως συχνά άλλωστε πράττει, προσπαθεί να συνδυάσει δύο πράγματα. Μιλά για την απαγόρευση του short selling των ανοιχτών πολίσεων. είτε για τα κυρίαρχα ε, τα συμβάσεις δηλαδή τη στάθμισης ψωτικού κινδύνου ή για κάποια άλλα εργαλεία, λέγοντας ότι ε, τελικά δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία μπορούσαν να επιληθούν. Και λέει στην αιτιολογική έκθεση ότι είχε ζητήσει από μια ομάδα γνωμόνων ε, στις κινητές αξίες, την ομάδα ΕΣΜΕ, μια ανεξάρτητη κατά Κομισιόν Επιτροπή, η οποία θα παρήχε συμβουλές και η οποία απαρτιζόταν από συμμετέχοντες στην αγορά. Δεν ξέρω, αυτοί που βοηθούν την Επιτροπή να συντάσει τις προτάσεις οδηγίας ή κανονισμού, γιατί εδώ πρόκειται περί ε, σχεδίου κανονισμού υπάρχουν κάποιοι εμπειρογνώμονε. έχω τον κατάλογο, είναι 20 τον αριθμό, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και όλοι προέρχονται από τη βιομηχανία. Όλοι. Κανείς δεν είναι ακαδημαϊκός, ούτε προέρχεται από κάποιον άλλο κλάδο. Είναι βέβαια όλοι οι υπέρμαχοι των επιχειρήσεων, από τον κλάδο δηλαδή από τον οποίο προέρχονται. Και ανοίγω μια παρένθεση. Πρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου Μπαρνιέ που ζήτησε από τις υπηρεσίες του στο μέλλον η ομάδα που παρέχει συμβουλές να μην, εκπροσω... να μην απαρτίζεται μόνο από επιχειρηματίες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρήσεων. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τις ε, συμβάσεις αντιστάθμισης πιστοτικού κινδύνου συγκεκριμένα, μοιάζουν με ένα ασφάλισης. Αλλά ασφάλεια λίγο περίεργη, λίγο ιδιαίτερη. Γιατί αυτοί που συνάπτουν αυτού του είδους τις ασφάλειες, αυτούς τις ασφαλίσεις, ουσιαστικά δεν είναι σίγουρο το κατά πόσον καλύπτονται, γιατί δεν εκτίθενται ουσιαστικά σε κάποιο ανοιχτό κίνδυνο. Οι συμβάσεις αυτές αντιστάθμιση συνήθως είναι ένα είδος στοιχήματος και έχουν και ένα χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Και το είδαμε αυτό. Στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης είδαμε αστρονομικά ποσά. Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το παγκόσμιο ΕΠ. Και το ποσό των συμβάσεων αντιπροσώπευε το δεκαπλάσιο των απολειών που υποτίθεται ότι θα κάλυπτε. Άρα ουσιαστικά δεκαπλασίασαν τους πραγματικούς κινδύνους που προϋπήρχαν της δημιουργίας τους, τα CDS αυτά. Δημιούργησαν ένα πραγματικό τέρας λοιπόν. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφέρω έναν Άγγλο συγγραφέα και αν δεν ακούτε αγγλικά καλό θα ήταν ίσως ε, να βάλετε τα ακουστικά σας, αν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα του Σέξπιρ. Λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουμε ακόμη τα CDS ε, γιατί μια, μια ανοιχτή πώληση σημαίνει ότι παίρνουμε την ασφάλεια για ένα ομόλογο που δεν έχουμε στην κατοχή μας. Ή ουσιαστικά πρόκειται για ένα στίχημα, για κερδοσκοπία. Δεν έχει κανένα κοινωνικό ούτε οικονομικό όφελος. Ιδίως γιατί ανοιχτέ πωλήσει σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς ε, να τις ταυτίσει με ληστεία τράπεζας. μπορεί κανείς τελικά να εξασφαλίσει και να ασφαλίσει μόνο αυτό το οποίο έχει στην κατοχή του. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε απλά για στοίχημα, αλλά μιλάμε για ένα μέσο που επιτρέπει στον πολίτη να μειώσει τους κινδύνους του. Δεν είναι αριστεριστής αυτός ε, που τα ε, λέει αυτά, αλλά είναι ένας από τους πιο σεβαστούς ε, αναλυτές των Financial Times και θα μπορούσα να πω κι άλλα και να διαβάσω κι άλλα σχετικά. Νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε. Πάντως, κάποιες πρακτικές της αγοράς για μένα είναι προφανές ότι δεν έχουν μπορούν να έχουν καμίας υποστήριξης. και δεν γνωρίζω κανέναν οικονομικό κλάδο που κάποιος μπορεί να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει, μόνο το ναι short selling. Είναι το μόνο πράγμα που, που ξέρω. αν προσπαθήσει κανείς να πουλήσει ένα αυτοκίνητο που δεν έχει, που δεν είναι δικό του, θα πάει στη φυλακή. Αλλά στον τομέα των οικονομικών μπορεί να κάνει κανεί ό,τι θέλει. Πάντω είδαμε ιδίως μετά από αυτή την κρίση στο διεθνές επίπεδο, που δεν έχει λήξει ακόμη, και αν κατατύχει πληγή ρευστότητα και υπάρξει μεγαλύτερη διακύμανση στις ε, αγορές, θα σας πω εγώ ωραία. Και λοιπόν, και τι έγινε. Γιατί αυτή η διακύμανση ίσως παροτρύνει κάποιους κερδοσκόπους να γίνουν πιο σόφρονες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα τόσο ωραίο να ακούει κανείς τον, ως αγορητή τον Ρόμπερτ Γκέμπερς. Καμιά φορά διαρωτάται κανείς αν ήταν υπουργό στο Λουξεμβούργο ή τέλος πάντων όταν ήμουν εγώ στο κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη πάντα ανησυχούσαμε σε σχέση με χρήματα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ε, τι συνέβαινε. Δεν ανησυχούμε, ε, δεν είχαμε κάποια ανησυχία διότι ξέραμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ανοιχτών αγορών και τελικά υπήρξε δυνατότητα να επιβιώσουμε σε σχέση με τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις επί δεκαετίες αυτό έκαναν και εμεί δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν να είμαστε επιθετικοί υπό... ω φιλελεύθεροι, διότι ακριβώ τι ίδιε απόψει ε, είχαν. Ο Τζορτ Σόρο τώρα, αυτό ο σημερινό ήρωα, κερδοσκοπούσε, καθώ γνωρίζετε. Κερδοσκοπούσε κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Έγινε δισεκατομμυριούχος, τώρα μπορεί να καταρτίζει τους κανόνες και κανονισμούς. Ήταν κακό αυτό για την χώρα μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την επιτροπή στην οποία ε, βρισκόμουν 500% επιτόκιο είχαμε χάθηκαν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης είχαμε τεράστια ε, επιτόκια αλλά αυτά Ρόμπερτ αυτά ήταν το βάθρο για την να, αλλάξει, η χώρα μας, να υπάρξει αλλαγή. Και τώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει, διότι λόγω αυτών που συνέβησαν τη δεκαετία του 90, εμείς στη Σουηδία σε καλύτερη θέση από ό,τι οι άλλοι. Είναι πάντα λοιπόν κακό αν κάποιο αποκαλύπτει πόσο αδίστακτη είναι η συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου. Δεν είμαι τόσο βέβαιο γι' αυτό. Όμω σίγουρα θα πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρξαν πολλά, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και αυτό αναφέρεται, αναφερόταν στην έκθεση της κυρίας Μπερές και υπερψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία αυτό ότι δεν ήταν ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο οποίο φιλόταν αυτό μία αιτία και μόνο. Ναι, καμιά φορά πρέπει να το αναφέρουμε σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ήταν ένα συνονθήλευμα, ένα σύνολο διαφορετικών συντελεστών και παραμέτρων. Και οι πολιτικοί στην Ευρώπη και εκείνοι πρέπει να υπομισθούν. Επομίζονται ευθύνε για αυτή την κατάσταση πραγμάτων τότε. Λοιπόν, κύριε Κομφέν, πιστεύω ότι στο τέλο και πρέπει να το πω αυτό ότι στο τέλος ε, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όμως στο τέλος. Στην αρχή όμως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θέματα που θα προταθούν σε σχέση με τροπολογίες. Στο τέλος όμως πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αν καταλαβαίνω σωστά όσα αναφέρθηκαν, αναφέρθηκε από τον Μάρκο τα χρειαζόμαστε, λέει όλα αυτά. Αν κατάλαβα σωστά εννοεί αν χρειαζόμαστε το short selling ή όχι. Αυτό όμω πρέπει να το αποφασίσει η ίδια η αγορά, δεν το αποφασίσουμε εμεί. Εντάξει. Ναι, μα γι' αυτό είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Γι' αυτό με έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι να πω, να πω ότι δέχομαι όλα τα δικά σου επιχειρήματα. Αυτό θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση τότε και πολύ βαρετή η συζήτηση που θα είχαμε. Πρέπει να μου δώσεις το δικαίωμα να εκφράζω τις απόψεις μου με αυτόν τον τρόπο. Η δική μου πείρα από τη δική μου χώρα αποδεικνύει ότι τα πράγματα είχαν έτσι όπως τα παρουσιάζω. Καμιά φορά πρέπει να ρωτήσεις εσύ του σοσιαλδημοκράτες εταίρους σου, ε, συντρόφους σου, τι έγινε, τι έγιναν αυτά τα τελευταία χρόνια. Ερώτηση, χρειαζόμαστε λέει αυτό το νομοθετικό έργο, αυτό το νόμο. Αυτό είναι υπόθεση ε, αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το απαντήσει. Αυτό είναι το οποίο ρωτάνε οι πολίτες, ζητούν οι πολίτες της Ευρώπης. Πόσες φορές ε, απευθύνεται το, το ζήτημα από τους πολίτες θέλουμε να απαγορευτεί το short selling και γιατί δεν το κάνετε. Ναι, εντάξει, κάθε μέρα ίσως εσείς το λαμβάνετε. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει. Και τότε θα πρέπει φυσικά να εξετάσουμε και κάτι άλλο. Αν είναι κακό, αρνητικό αυτό, ή είναι κακό, είναι αρνητικό για μια λειτουργούσα αγορά, κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν ήταν κακό στη δική μου χώρα και δεν μπορούμε διαρκώς να κάνουμε εξαιρέσεις και να λέμε ότι είναι διαρκώς κάποια εξαίρεση. Όταν η κρίση ήταν τόσο κακή, είχε φτάσει σε τόσο αρνητική κατάσταση, δεν το απαγόρευσε η κυβέρνησή μα. Όμω η γερμανική κυβέρνηση το απαγόρευσε. Το απαγόρευσε κύριε, το απαγόρευσε. Δημιουργούσε προβλήματα. Ιδιαίτερα δημιουργούσε προβλήματα σε μικρέ αγορέ μικρών χωρών. Ίσως όμω δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό, δεν σα νοιάζει. Κι όμω ήταν βλαπτικό για αυτέ. Και θα πρέπει να υπάρξει κάποιο εναρμονισμό όσον αφορά την νομοθεσία. Συμφωνώ για το εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο να εξετάσουμε διαφορετικέ προτάσεις επίσης. Είμαι πρόθυμος να ακούσω ποιε είναι αυτές. Όμως κύριε Γκέμπερ και κύριε Κομφέν και ίσω και εσύ ο ίδιο Μάρκους Φέρμπερ, εσείς πρέπει να μας υποβάλλετε κάποια αποδεικτικά στοιχεία ναι, μην το λέτε έτσι ως θέσφατα, διότι εγώ ρωτούσα και ζητούσα, δώστε μας κάποια παραδείγματα που να δείχνουν ότι το short selling ήταν αρνητικό. Αποδείξτε το, δώστε κάποια τεκμήρια, δώστε συγκεκριμένα χειροπιαστά παραδείγματα. σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Απαντά, όχι, αυτό δεν ήταν απλό short selling, naked short selling, ήταν ένα συνδυασμός ο Μπάνι Φρανκ ήταν εκείνο που το είπε σε σχέση με Φρέντι Μάρκ ότι θα έπρεπε να δίνονται λέει δάνεια σε όλου. ακόμα και σε εκείνου που δεν μπορούσαν να τα ξεπληρώσουν και μετά υπήρξε αυτό το πατατράκ πρέπει να το δει κανεί στι ρίζε του αυτό και να υπάρχουν κανόνε. είναι λοιπόν καλό ή όχι για την αγορά το short selling εγώ από την προσωπική μου πείρα πρέπει να πω και για την αγορά στη χώρα μου ότι θεωρείται ότι είναι καλό και ότι θα μπορούσε ουσιαστικά να παρακολύσει την αγορά στη λειτουργία της αν το απαγορέψουμε. Αλλά είμαι πρόθυμος να ακούσω αντίθετα επιχειρήματα. Και πάντα όταν λέγεται μεγαλύτερη διαφάνεια, συμφωνώ με αυτό πολύ καλά. Μεγαλύτερη διαφάνεια. Διαφάνεια λοιπόν. Μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα τιμών κατοφλίων επίσης. Μπορούμε επίσης να συζητήσουμε το θέμα καθορισμού επιμερισμού, flagging και όλα τα διαφορετικά αυτά συναφή θέματα. Αλλά μην λέμε εκ προημίου πρέπει να απαγορευτεί το short selling, τελεία και παύλα. Εκεί ολοκληρώνω και λέω εντάξει δώστε μας κάποια καλά πιστικά παραδείγματα. Το παράδειγμα των Lehman Brothers δεν είναι καλό, δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει κάποια χειροπιαστά παραδείγματα να μας δώσετε από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επαρκεί και δεν είναι καλό το αποδεικτικό στοιχείο για την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ζωντανή η παρέμβασή σας. Μας ε, δώσατε έτσι πιο πολύ και σε μας ε, ζωντάνια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάντοτε ε, είναι ωραίο να ακολουθεί κανείς την τα όσα είπαν οι Γκέμπελ και Σμιτ και να μπορεί να μιλήσει και αυτό στην ε, γλώσσα της λογικής. Εγώ νομίζω ότι έχουμε συνεργαστεί και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν ε, με τον κύριο ε, Γκέμπελς και ίσως και στο μέλλον θα μπορούσαμε να ξανασυνεργαστούμε. Τώρα, χαιρετίζω τις προτάσεις της Κομισιόν όταν συζητήσαμε και τις, ε, τη διαχείριση των κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων ήταν από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Ε, είδαμε και τα θέματα του short selling αλλά και τα αντιμετωπίσαμε σε οριζόντια βάση. Ε, αυτό είναι θετικό λοιπόν και ελπίζω να έχουμε χρόνο να κάνουμε και τις ερωτήσεις μας. Νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμητό αυτό. Ο Μάρκους έκανε τις δικές ερωτήσεις και όλοι θέλουμε απαντήσεις στις απορίες μας μία από τι ερωτήσει που θα μπορούσε να τεθεί είναι πρώτα απ' όλα να δούμε κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Ποια είναι τα θετικά των ανοιχτών πωλήσεων του short ε, ε, selling. Ρομπέρ, δεν κατάλαβα ακριβώ τι είπε. Είπε γιατί ε, κάποιο ε, θέλει να πουλήσει κάτι που δεν είναι στην κατοχή του. Μιλά για short selling ή για το naked short selling. Πολλοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι πουλούν πράγματα που δεν του ανήκουν, όπως παραδείγματο χάρη ναι, η εταιρεία Amazon ε, που κάνει short selling οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί που πουλούν κάποια ε, τα κτλ. Λοιπόν υπάρχουν πολλοί οποίοι πουλούν πράγματα τα οποία δεν τους ανήκουν. Για τη ρευστότητα είπες εσύ κάποια πράγματα, δεν συμφωνώ απόλυτα. αν κάποιες αγορές προβούν σε πολύ προσεκτικές αναλύσεις, νομίζω ότι μπορούν να, έχουν και κάποια κέρδη. Και είδαμε ότι πολλές φορές ε, το short selling σε πολλές περιπτώσεις, τα Icon Lehman Brothers, ε, ήταν ε, το θετικό στοιχείο και πολλές φορές βοηθά και το να μην δημιουργηθούν ε, φούσκες. Ένα από τα σημεία στα οποία μπορώ να συμφωνήσω ότι χρειάζεται είναι βελτίωση της διαφάνειας και ελπίζω οι ρυθμιστές να έχουν στη διάθεσή τους και τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους συστημικούς κινδύνους. Και όπως και όλοι, ρωτώ και εγώ, γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό. Και αν έχουμε κανονισμό, Πώς θα φροντίσουμε να μην ε, είναι ένας ε, που θα ισχύει για όλους. Όταν είχαμε πρωτομιλήσει για ε, τα, τα είχε πει και ο κύριος Γκοζές κάποια πράγματα και είναι διάφορες, οι μεγάλες οι διαφορές από τα equity funds για παράδειγμα. Θα ήθελα να ακούσω και τα επιχειρήματα και υπέρ και κατά. Κάποιες τυχές θέλω να διευκρινιστούν περισσότερο. Τι θα πει πρώτα απ' όλα naked short selling. Κάποιοι είναι υπέρ, κάποιοι θεωρούν ότι είναι χρήσιμος ε, κάποιοι είναι κατά, αλλά τι είναι. Και λέει, locating a reserve, reserve, απόθεμα. Τι απόθεμα είναι αυτό. Και μοιάζει με άλλες δικαιοδοσίες, ε, περιλαμβάνει ρευστότητα, κλείδωμα κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Τι είναι ακριβώς ή απλά είναι μια ρύθμιση, να υπάρχει μια ρύθμιση για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Τώρα, η δημοσιοποίηση στην κοινή γνώμη. Θα πρέπει να προσέξουμε πως υπάρξουν επιπτώσεις οποίες δεν θα επιθυμούσαμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε και καλά στην όλη, στον διάλογο που θα έχουμε. Αν κάποιο, παραδείγματο χάρη, ε, είναι ένα μικρό ερευνητικό οίκο που κάνει προσεκτική έρευνα και εντοπίσει κάποιε φουσκωμένε μετοχέ κατά κάποιο τρόπο, ε, τι πρέπει να κάνει, Πρέπει να την κοινοποιήσει την έρευνα αυτή σε όλου, ε, στου μεγάλου ερευνητικού οίκου. Και για τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Αρχή ΕΣΜΑ έχω επίση τις αμφιβολίες μου και τα ερωτηματικά μου. τι θα γίνει σε περίπτωση ανάγκης, σε έκτακτες περιστάσεις. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και για το flagging. Πόσο ακριβείς μπορεί να είναι οι πληροφορίες για το flagging και τι σχέση μπορεί να έχει και με το κόστος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, απορίες που έχω για τον κανόνα circuit breaker. Έγινα κάποια ε, πρόταση, αλλά θα πρέπει να αυτό το 10%. Αλλά τι γίνεται με κάποιες ε, μετοχές που έχουν μεγάλη διακύμανση. Και σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική αγορά ε, ταύσιν ημερών, θα έπρεπε να έχουμε κάποια στοιχεία υπάρχει πρόβλημα το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν υπάρξουν στοιχεία που το αποδεικνύουν, είμαι υπέρ, αλλά αλλιώ δεν έχει νόημα. Κάτι άλλο που με έχει προκαλέσει σύγχυση, όπω και στην συζήτηση που είχαμε προηγουμένω και με τα ε, MIFIDs, πάντα μιλάμε και για την απάτη. Αν γίνεται short selling, ε, δηλαδή με την διασπορά ε, φημών, ψευδών φημών, θα πρέπει να δούμε η υπερρύθμιση θα έχει κάποια αποτελέσματα. Ας ε, διατηρηθούμε και εμείς αυτό που ρωτά ο Μάρκο, αυτό που ρωτά ο Όλε. Και να δούμε τελικά ποιο μέρος των δραστηριοτήτων ε, αφορά αυτό. Και να δούμε και τι προβλήματα, αν υπάρχουν, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν πάντως να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς διαφάνειας και όχι υπερβολικών ρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ουσιαστικά ο σκιώδη εισηγητή μα για αυτή την έκθεση είναι ο Τόμα Έντλ. Όμω σήμερα δεν παρίσταται. Έχει άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει. Γι' αυτό με παρακάλεσε εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσει για, τον, για λογαριασμό του ανταυτού. Πρέπει, θέλω πρώτα στον Όλε Σμιτ να πω κάτι. Καταρχήν σωστό είναι ότι ζωγόνησε αυτό τη συζήτηση και αυτό δεν είναι αρνητικό το να έχει κάποιο διαφορετική άποψη από το να συμφωνούν όλοι με μια άποψη. Αναφέρθηκε ότι μέσω κάποιων διαδικασιών τη αγορά στη Σουηδία υπήρξαν κοινωνικέ αλλαγέ που επιβλήθηκαν. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματο. Είπατε όμω επίση ότι υπήρχαν πάνω από 100.000 ε, άνεργοι και αυτό είναι αναγκαίο. Να δούμε και αυτή τη συνιστόσα. Να δούμε για αυτού του ανθρώπου τι γίνεται για αυτού που έχασαν τη δουλειά του. Μέσα στο πλαίσιο τη κρίση καταλήξαμε άνθρωποι να έχουν χάσει τα δικαιώματα σύνταξή του, όσον αφορά τη συνταξιοδότησή τους με την, με την απώλεια των κεφαλαίων και με αυτά τα χρηματικά προϊόντα πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν μπορεί να πει κανεί η αγορά θα τα ρυθμίσει όλα και θα δώσει την απάντηση αν αυτά τα προϊόντα είναι αναγκαία στην αγορά ή όχι. Είμαι πεισμένο γι' αυτό γιατί διαφορετικά δεν θα συζητούσαμε αυτά τα θέματα. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για κοινωνική οικονομία της αγοράς και πίσω από αυτό βρίσκεται μάλλον και σίγουρα η αρχή ότι δεν μπορεί η αγορά να τα ρυθμίζει όλα αφεαυτής. Είναι πολιτική απόφαση να δούμε τι είναι σκόπιμο και χρήσιμο και τι όχι. Και σε σχέση με τις δικές μας απόψεις να λάβουμε υπόψη αυτά και να μεριμνήσουμε να μην χάνουν τη θέση εργασία του άνθρωποι. Άνθρωποι που δεκαετίες πλήρωναν τα, το μέρισμα στη, για την σύνταξή τους να μην χάνουν στο τέλος τέλος τη σύνταξή τους και μένουν γυμνοί. Αυτό είναι μια πολιτική πρόκληση σε σχέση με τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και καθήκον μας, στόχος που πρέπει να επιτελεστεί και θέλω να το υπογράψω σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε και θα υποστηρίξουμε τον εισηγητή να διασφαλιστεί αυτή η πτυχή. Και αυτά που είπε ο Ρομπέρ δεν είναι λανθασμένα, δεν, είναι, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως έναυσμα να ε, διαφωνήσει κανείς με αυτά και πρέπει να δει κανείς και για τους σοσιαλδημοκράτες ότι είχαν και διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Δεν πρέπει εδώ να κάνουμε υπέρβαση του παρελθόντος και απολογισμό λαθών, αλλά να δούμε τι καλό μπορούμε να κάνουμε και να πορευτούμε προς μια κατεύθυνση και αυτό θα είναι καλό. Ένα πράγμα θέλω να πω. Γυμνές πωλήσει, ε, naked short selling. Ναι, ε, σίγουρα σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Να δούμε τι κάνει η κυρία Μέρκελ τώρα με αυτό θα μπορούσε κάτι άλλο να κάνει και δεν το κάνει. Ναι, τέλος πάντων, πάλι σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει, α μην κάνουμε γερμανογερμανική συζήτηση εδώ, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπό το δικό μα πρίσμα γυμνέ τέτοιε πωλήσει είναι απλή κερδοσκοπία. Γυμνή κερδοσκοπία. Και δεν βρίσκουμε κανένα λόγο να μπορέσουμε να καλύψουμε κάτι και να το δεχτούμε. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε, σύμφωνα με τι δικέ μου γνώσει, να δούμε τι γίνεται με τον όγκο και με την διασφάλιση της δυνατότητας ε, και μάλιστα σε τέτοιο όγκο πολλαπλάσιο του αμερικανικού προϋπολογισμού. Δηλαδή εδώ έχουμε μια τεράστια κερδοσκοπική φούσκα που δημιουργείται και που στο τέλος θα ήθελα να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, αλλά φαίνεται ότι δεν την έχουμε τελείως ξεπεράσει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση του τομέα. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Αυτό υποστηρίζουμε. Αυτό το αίτημα που ο Πασκάλ είχε διατυπώσει και αυτό θέλω εγώ να πω ρητά και κατηγορηματικά. Αυτό υποστηρίζουμε. Σε διαβούλευση φυσικά με τον εισηγητή θα συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ για την προσοχή. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω αμφιβολία ότι με την τεχνογνωσία και την πολιτική αντίληψη του Πασκάλ θα κάνουμε καλή δουλειά εδώ. Να υπογραμμίσω όμως ότι ο Μάρκος έθεσε τα σωστά ερωτηματικά και ήδη έχουμε μια έτσι, γεύση απάντησης. Καταρχήν, στο, πολιτικό, στο πολιτικό μας κόσμο μιλάμε για κοινωνική οικονομία της αγοράς και το κοινωνική δεν το λέμε τυχαία. Να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Και το θέμα του ποια είναι η θέση της αγοράς και ποια κομμάτια της αγοράς θα πρέπει να ρυθμίζονται αποτελεί ένα ουσιώδη ζήτημα σήμερα. Νομίζω ότι εθελοτυφλούμε αν δεν δούμε τις επιπτώσεις της κρίσης που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε τα θέματα της ασφάλειας εργασίας. Δεν γίνεται όμως να θεωρήσουμε ότι έχει περάσει καταιγίδα και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Και δεν χρειάζεται βέβαια να επιστρέφουμε σε ιδιαίτερα τεχνικά ζητήματα. Αν μου επιτρέπετε να συνάξω τα συμπεράσματα από αυτό που θα ψηφίσει την Πέμπτη το Κοινοβούλιο του IFM, Είχαμε 200 συναντήσει με του λομπίστε και τη μηχανία και μετά πολλού μήνε ε, συνομιλιών έχω την εντύπωση ότι τώρα πια έχουμε μια πολιτική θέση. Δεν χρειάζεται να επισέλθουμε στις λεπτομέρειε του κανονισμού αν δεν ξέρουμε ακριβώ ποιοι είναι οι στόχοι μα. Οι απότεροι μας στόχοι. Και στο Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θα πρέπει να καθορίσουμε αυτού του στόχου και να προσπαθούμε να τους πετύχουμε ανεξάρτητα από το επίπεδο λεπτομέρειας του κανονισμού. Κύριε Σμιτ, να σας πω ότι εγώ τους πολίτες του συναντώ κάθε Κυριακό στην Ορμανδία που είναι η περιφερειά μου και τα ερωτήματα αυτά μου τα θέτουν οι ίδιοι οι πολίτες οι γεωργοί οι βιοτέχνε, οι εργάτε θέλουν αυτά τα ερωτήματα. Βεβαίω δεν επισέρχονται στα τεχνικά ζητήματα του short selling. Μου λένε όμω, τι κάνετε εσεί στην Ευρώπη για να αποφύγετε την επανάληψη τη κρίση. Τι κάνετε στην Ευρώπη για να μην υπάρχουν ε, παράδοξες καταστάσεις ή απαράδεκτες, μη αξιοπρεπείς. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, αυτό θα πρέπει να δούμε. Όπως είπε και ο Σμπαρνιέ, έχουμε το πλαίσιο έχουμε τη βάση. Τώρα θα πρέπει να αρχίζουμε να χτίζουμε το IFM πρώτα. Είδαμε και με τι δυσκολίε, γιατί όπω έλεγε και ο Ρομπέρ προηγουμένω, πίσω από αυτά τα ζητήματα δεν κρύβονται τα ζητήματα τη εθνική κυριαρχία και η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με εθνικέ αρχέ, όπω έλεγε ο, ο Βέλγο Πρόεδρευμα πρόσφατα. Ε, έχουμε να κάνουμε τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία τη οικονομία. Κανεί δεν είπε ότι η χρηματοοικονομική βιομηχανία θα πρέπει να καταστραφεί. Θα πρέπει όμω να τηρήσει τον δικό τη το στόχο, δηλαδή να βοηθήσει τη λειτουργία τη οικονομία, να προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εδώ λοιπόν αυτό θα μπορούσε να ήταν απάντηση στα πολιτικά ερωτήματα που θέτει ο Μάρκος μέχρι που θα πάμε και αν το έχουμε κάνει αυτό τότε θα έχουμε κάνει την δουλειά μας ως ε, βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κάριντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω ένα σχόλιο. Συζητιέται πολύ η καθαρά κερδοσκοπική φύση του Νέκη Short Selling. Εγώ είμαι από τη Λετωνία όπου 50 χρόνια έλεγαν στις αρχές πόσο κακή είναι η κερδοσκοπία αυτό μου ακούγεται λίγο παράξενο η κερδοσκοπία είναι παντού γύρω μας. Αν έχει επενδύσει κανεί σε ένα ιδιωτικό σε ταμείο, κερδοσκοπεί. Τι θα κάνουν λοιπόν οι διαχειριστέ του ταμείου για να το κάνουν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Οι αγρότες, όπως αναφέρθηκε προηγουμένω, προηγουμένως, κερδοσκοπούν με τις καλλιέργειέ τους την κατάσταση του εδάφου ώστε να βρουν τι κατάλληλε καλλιέργειες που θα καθορίσουν τέλο πάντων τι τιμέ. Τη εισοδία τα επόμενα χρόνια. Όλοι λοιπόν κερδοσκοπούμε συνέχεια. Και νομίζω ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην κερδοσκοπία και στο κακό naked short selling λόγω τη κερδοσκοπία, επειδή θα έλεγα τότε ότι πηγαίνουμε σε νερά. Νομίζω ότι αυτό πρώτον είναι διάφοροι είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο συστημικό πρόβλημα, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, το τι επιπτώσει έχει τον έγκυο selling στις αγορές. Και αν θεσπίσουμε κανονισμό, τι θα αντιμετωπίζει. Όχι το γεγονό ότι υπάρχει χειροδοσκοπία. Ε, τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να απαγορεύσουμε και τη γεωργία, επειδή είναι κακή πρακτική και δεν έχει καμία κοινωνική αξία. Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα γιατί κάποιε δραστηριότητε έχουν ε, κοινωνικά στοιχεία, άλλε όχι, φαίνονται λίγο παράξενα. Θα πρέπει όμω να πούμε και να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συστημικές επιπτώσεις και αν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες ή αν αντίθετα κατηγορούμε κάτι επειδή οι ψηφοφόροι μας ανακάλυψαν το κακό short selling, τον negative short selling Οπότε θα πρέπει να το χτυπήσουμε και να το απογορεύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να τα υπολογίζουμε όλα αυτά. Εγώ δεν θα ακολουθήσω κάποια συγκεκριμένη πλευρά σε αυτή την επιχειρηματολογία. Θα πρέπει όμως να το δούμε ξεχωριστά και να το απομακρύνουμε από αυτές τις συναισθηματικές συζητήσεις για την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ βάλω τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών πριν την Κομισιόν και τον εισηγητή. Εγώ χαιρετίζω αυτό που είπε ο εισηγητή ότι θα κοιτάξει το θέμα με τρόπο έξυπνο και θα, εξηγήσει, θα εξετάσει τα γεγονότα. Να δει δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν τρόποι εποπτείας ή ελέγχου. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην οδηγία AMF, AIMF. Οι χώρες που ανησυχούν για τα hedge funds είναι αυτές που δεν έχουν κανόνες για τον έλεγχο των hedge funds που έρχονται σε άμεση επαφή με τους επενδυτές. Αυτές οι χώρες λοιπόν που ανησυχούν με την αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων είναι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν συστήματα κοινοποίηση στοιχείων αυτών των συναλλαγών προς, τους, προς το κοινό. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιους κινδύνους. Πριν λοιπόν βιαστούμε και κάνουμε κάτι το άσχημο, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει, τι προϋπάρχει μάλλον, και να μην μπερδέψουμε ότι είναι βλαβερό με ό,τι κάνει καλό στην αγορά. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε και να διηγήσουμε στην αφαίρεση δραστηριότητες από την αγορά επειδή δεν μας αρέσει και να είμαστε τόσο αυστηροί. Όπως είπαν κάποιοι, το short selling είναι ένας τρόπος με τον οποίο επιβίωσαν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Ένα τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το εξή. Τα naked CDS. Θέμα που συζητήσαμε προηγουμένω στο πλαίσιο των παραγόγων στην Επιτροπή μα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγοράζουν τα CDS και έχουν πραγματικό γνήσιο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη χώρα και όχι στο ομόλογο αυτό καθευτό. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Μπορεί να υπάρχει ας πούμε ένα είδος ε, δίκτυ παραγόγων. Αλλά νομίζω ότι είναι κανείς αλλού ότι αν ότι θα αλλάξουν οι τιμές αυτών των παραγόγων και ότι θα μπορέσουμε τέλος πάντων να διαχωρίσουμε το ενδιαφέρον κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ε, ενδιαφέρον ας πούμε, για τις διακοπές τους σε μια χώρα και με αυτό των ανθρώπων που έχουν ενδιαφέρον για την τιμή του παραγόγου ή την τιμή του ομολόγου. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αν οι αγορές θεωρούν ότι μια χώρα ε, είναι άτακτη, το θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας τρόπος κάλυψης του κινδύνου των παραγόντων της αγοράς. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο συμφέρον στην ανέκη της CDS να εξετάζουμε κατά πότε αφορά το ομόλογο αυτό καθεαυτό. Επειδή θα είναι δύσκολο να διακρίνουμε εκεί τι είναι νόμιμο και ηθικό και να το τεκμηριώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν πριν προχωρήσουμε σε απαγορεύσει, θα πρέπει να κάνουμε και εμεί τη δουλειά μα, να μελετήσουμε, να δούμε πόσο και χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο και να πω ότι για τα naked CDS έχουμε στοιχεία από τα διάφορα μητρώα. Πάρα πολλοί αντίδρασαν και είχαμε και αναφορές στον τύπο κάπως ε, οξύες. Η ε, κυρία Βαλέντσα. Ευχαριστώ πολύ. Με ικανοποίησε πάρα πολύ το γεγονός ότι η πρόταση της Κομισιόν προκάλεσε τέτοια συζήτηση ε, στην Επιτροπή σας. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο, πώς προέκυψε η πρόταση. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν μια πρόχειρη ούτε βιαστική αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκίνησε η συζήτηση όπως γνωρίζετε το 2008 και εμείς ζητούσαμε από τους νομοθέτες να καταλήξουν σε μια κοινή λύση γιατί ε, υπήρχε τα περιθώρια για ρυθμιστικά και είχαμε και κάποια μνήματα από τις αγορές ενώ ταυτόχρονα σε άλλες ε, δικαιοδοσίες ιδίως της ΕΠΑ ε, γινόντουσαν προτάσεις για πιο δραστικά μέτρα. Άρα δεν είναι καινούρια η συζήτηση. Σίγουρα εντάθηκε η συζήτηση την τελευταία, την άνοιξη συγκεκριμένα και συμφωνώ με ορισμένους που είπαν ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερος ε, κακή όχι μόνο για μικρές χώρες αλλά και για μεγάλες χώρες γιατί υπήρχαν κάποια τοξικά προϊόντα διασπαρτά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε λοιπόν ε, ίσως κάποια μεγάλα κράτη-μέλη έκαναν ε, κάποιες ε, είχαν κάποιες πρόχειρες αντιδράσεις, κάποια κακά σχόλια ακούσαμε από κάποια άλλα κράτη-μέλη κτλ. Έτσι θελήσαμε εμείς να εκπονήσουμε αυτόν τον κανονισμό και βέβαια λάβαμε υπόψη και την Επιτροπή των Ευρωπαίων Ρυθμιστικών Αρχών και από την ΕΣΜΑ βέβαια. Ακούσαμε, υπόψη ακαδημαϊκές μελέτες και έγινε και μια δημόσια διαβούλευση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων ε, έως πέντε μηνών το πολύ. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο δεν είναι τη στιγμή, έχει ξεκινήσει πιο παλιά. Ξέρουμε ότι έχει επίγοντα χαρακτήρα αυτό το ζήτημα. Θέλουμε και εμείς να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς τα έξω για το πώς έχει κατάσταση στις αγορές. Ε, το δεύτερο ερώτημα, το χρειαζόμαστε τον κανονισμό αυτό. Η απάντηση είναι πάνω από καταφατική. Φυσικά και τον χρειαζόμαστε. Αν δει κανεί τις ε, προτάσεις, ε, έχει τρία σκέλη ο κανονισμός αυτός. Πρώτον, διαφάνεια. Δεύτερον, δίκτυα ασφαλείας. Τρίτον, έκτακτης, ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, και θα τα εξετηγήσω ένα-ένα. Διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι σίγουρα πάνω από απαραίτητη θα έλεγα εγώ. Ξεκινήσαμε τι συζητήσει με τους ε, ρυθμιστές και τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη συζήτηση αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα Έχουμε στοιχεία για το τι συμβαίνει στι αγορέ, γιατί δεν έχουμε. Και δεύτερον, μπορούμε να προχωρήσουμε αφού δεν έχουμε στοιχεία. Άρα λοιπόν κάπω έπρεπε να προχωρήσουμε και έπρεπε να δοθούν ε, εργαλεία για τη συλλογή στοιχείων, αποδεικτικών στοιχείων. Ταυτόχρονα θεωρήσαμε ότι δεν είναι καλή σταδιακή προσέγγιση, αλλά ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια πλήρη πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν Εισαγάγαμε αυτό το δίκτυο ασφαλείας, την ασφαλιστική δικλίδα και για να μην υπάρξουν ασυντόνιστες δράσεις, ούτε μονομερείς απαγορεύσεις, ε, εισαγάγαμε την ε, διαδικασία του κατεμπήγοντος έχοντας αυτά τα λεγόμενα circuit breakers έχουμε επίσης ε, πρόσθετη κοινολόγηση. Έχουμε και τα εταιρικά CDS. Μπορεί να ζητηθεί λοιπόν δημοσιοποίηση στοιχείων για τα CDS αυτά και κυρίως θέλαμε ένα σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Αρχή, την ΕΣΜΑ. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα συντονισμού στην ΕΣΜΑ και αν δεν υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να ε, δρουν μονομερώς, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι θέμα επικουρικότητας. Χρειάζεται συντονισμός, γιατί έχουμε εσωτερική αγορά. Ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θέμα. Αν έχει ισορροπία, τη σωστή ισορροπία η πρόταση, ήταν το τρίτο ερώτημα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα βασικά μηνύματα και τις βασικές διατάξεις, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα κατόφλια ή το flagging, όπως είδατε ίσως, ε, τα κατόφλια τα κατώτατα όρια είναι αυτά τα οποία θεώρησαν ε, ω κρίσιμα οι ίδιοι οι ρυθμιστέ και θεώρησαν ότι είναι τα καλύτερα, οι καλύτεροι ε, στην καλύτερη θέση για να μα δώσουν ε, τα στοιχεία. Αν όμω μπορούμε να έχουμε καλύτερα στοιχεία, βεβαίω μπορούμε και να αλλάξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναφορά το ίδιο, το ίδιο και σε ό,τι αφορά άλλου όρου για την ενεργοποίηση του κανονισμού. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Για να ολοκληρώσουμε θα δώσω τώρα τον λόγο στον Πασκάλ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές οι οποίοι ανέφεραν ορισμένα σημεία, τα οποία από ιδιαίτερο τεχνικά ε, ήταν ε, και μέχρι φιλοσοφικού ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Να προσθέσω κάτι που είχα ξεχάσει να αναφέρω στην αρχική μου παρέμβαση σε ό,τι αφορά το market maker είναι ένα και από τα σημαντικά που διακυβεύονται σε αυτό το κείμενο. Δηλαδή, μέσω ενός ε, ευρέως ορισμού για το market making, κάποιοι ε, φορείς θα μπορούσαν ενδεχομένως ε, να κάνουν κάποιες συναλλαγές, να προβούν σε κάποιες πράξεις και να έχουμε στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ αυτών τα οποία εξαιρούνται στο market maker, αλλά στην ομπρέλα, στην ομπρέλα, κάτω από την ομπρέλα market maker γίνονται κάποιοι ε, και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός ορισμός του όρου, της έννοιας για να μην υπάρχει εστρέβλος του ανταγωνισμού. Το marketing επίσης αναφέρθηκε και από τον Μάρκους και από άλλους. Το άρθρο της Κομισιόν για αυτό το θέμα είναι σημαντικό και νομίζω ότι είναι μόνο 4-5 γραμμές, ε, είναι μικρό. Άρα καλό θα ήταν να το διευκρινίσουν περισσότερο. Σε τι θα χρησιμεύσει, πού θα σταλεί, υπό ποιες όρους κτλ. Υπάρχουν νομίζω πρακτικές πληροφορίες που πρέπει να προσθεθούν. Και το τελευταίο, για τον Όλε Σμιτ φυσικά, κάθε φορά εκπλήσωμαι όταν ακούω τους φιλελεύθερους να ε, μιλούν κατά της διαφάνειας. Ποιος είναι αυτός που ωφελείται από το naked ναι short selling. Δείτε ε, ποιος ε, ωφελείται σε βάρος ποιου. Έχουμε ε, τους βραχυχρόνιους που ωφελούνται κατά των μακροχρόνιων. Εγώ δεν θέλω όμως ε, να υποφελούνται μόνο αυτοί, αλλά θέλω και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αποταμιεύσεις μακροπρόθεσμα επίσης να ωφελούνται. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Η εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα είναι 13 Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο ε, θα συζητήσουμε, 1η Φεβρουαρίου ε, θα δούμε τις τροπολογίες ε, και θα ψηφίσουμε στις 7 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Και μετά κάποια στιγμή στην Ολομέλεια θα πάει η έκθεση. Ο εισηγητής συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα περνάμε στο σημείο 5 της μερισιάς διάταξης. Έχουμε και τους 20 αξιολόγησης, αλλά στο τέλος, πενθυμίζω, Πρώτα απ' όλα όμως θα δούμε την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που την χάνουν δημόσιας στήριξης. Ο Άρτουρς, ο οποίος μιλάει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να λάβει το λόγο. Είναι απασχολημένος βέβαια αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ σαγέτη χρειάζομαι τον Άρτουρς να μας παρουσιάσει την έκθεσή του, τη γνωμοδότησή του. Είμαστε στο 5, συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τα καλά μαντάτα για αυτή την έκθεση είναι ότι έχουμε 13 τροπολογίες όλες και όλες. Θα προσπαθήσω λοιπόν πολύ σύντομα, χωρίς να επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες, να πω ότι πιστεύω ότι για την τροπολογία 4, 5 και 8 αυτές οι τρεις τροπολογίες είναι πανομοιότυπες στην κατεύθυνσή τους. Λένε ουσιαστικά ότι όταν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ε, υπηρεσιών πιστώσεων για τις εξαγωγές τους ε, εργάζονται με κάποιο τρόπο πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική τροπολογία να καλυφθούν αυτές οι τρεις. Η τροπολογία 5, ουσιαστικά, συγγνώμη, η τροπολογία 7 στη συνέχεια ουσιαστικά αναδιατυπώνει με την μορφή που έχει πάρει του κυρίου Μπέρμαν τις γενικές θέσεις ε, που έχει λάβει αυτή η συμφωνία. Δεν το βρίσκω να είναι αυτό σε κάποια αντίφαση και μπορεί να υποστηριχθεί ως αίτημα. Η τροπολογία ζητεί από το Συμβούλιο ετήσια να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή, την λειτουργία και εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι κάποια αντίφαση λοιπόν αυτό, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Περνάμε στι 10, 11, 12 και 13 τροπολογίε που είναι παράλληλε προτάσει από τον κύριο Τρεμόσα και τον κύριο Άλβεσα από την Άλντε και τους Πράσινους. Και οι δύο ζητούν και αυτό συσχετίζεται με την διαφάνεια και τα μέτρα, πρόσθετα μέτρα για τη διαφάνεια στο παράτημα 1 λένε ότι το παράτημα 1 θα πρέπει να αναφέρει την χρήση των μέσων όσον αφορά το, τους ε, ε, ισολογισμούς για πλήρη διαφάνεια. Αυτό σε σχέση με την συζήτηση για τη διαφάνεια δεν βρίσκω γιατί δεν θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε ως αίτημα. Μπορούμε λοιπόν να το υποστηρίξουμε. Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Λάμπερτς. Προτείνει όχι μόνο αυτό, αλλά και δεύτερον οι εταιρείε είναι η τροπολογία 12 που υποφελούνται από πιστώσεις για τις εξαγωγές θα πρέπει να αναφέρονται αναχώρα πώς λειτουργούν αυτές οι πιστώσεις για τις εξαγωγές. Ανησυχώ για το κόστος αυτής της πρότασης κάπως πρέπει να πω και έχω κάποιες επιφυλάξεις για την υποστήριξη. Τώρα, κατά τα άλλα μπορούμε να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες και θα συνιστούσα να υπερψηφιστούν αυτές οι προτάσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 12 όμως έχω επιφυλάξεις, δεν είμαι υπέρ. Ευχαριστώ. Fine. Um... Um, Ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Ευχαριστώ την εισηγητή για τα σχόλια. καθυστιαστικά σχόλια. Κατανοώ την ανεργία που έχει στην ρύθμιση και στους φραγμούς προς την αγορά. Κατανοώ και εγώ γιατί είχα ίδια εμπειρία από τη Σοβιτική Ένωση όλα αυτά και αγορέ. και η και αξιολόγηση χρειάζονται κανόνες, οπότε έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι για αυτά τα θέματα σε συνδυασμό με τους στόχους της Ένωσης και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια εύκολη λύση αύριο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Σταμόν. Ευχαριστώ κύριε Σικλούνα ένα λεπτό να πω ότι συμφωνώ με την άποψη του συγητή, δηλαδή ότι είμαστε σε καλή θέση για να βρούμε ένα συμβασμό μεταξύ όλων των ομάδων και θα έλεγα επίσης ότι στην τροπολογία 12 Lamberts στο δεύτερο σημείο θα προσθέσω ότι μόνο μεγάλες εταιρείες θα έπρεπε να δημοσιεύουν ισολογισμούς αναχώρα για να μην δημιουργήσουμε γραφειοκρατικό φόρτο στις μικρομεσαίες. Ο Φίλιπ δεν είναι εδώ, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνούσε με αυτή την πρόταση να μην προσθέσουμε δηλαδή γραφειοκρατικό κόστος στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Από την άποψη αυτή η διαφάνεια θα είναι υπέρ των επιχειρήσεων αν εμείς δηλαδή επιδείξουμε ευελιξία και πούμε ότι είναι αποκλειστικά το κόστος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για την τροπολογία 4, Γιούργεν Κλούτε, ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε την ορολογία εδώ. Επειδή αυτός χρησιμοποιεί το ρήμα shall στα αγγλικά. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να βρούμε μια άλλη διατύπωση να πούμε taking into account, να λάβουμε υπόψη δηλαδή τις αξίες και τις προδιαγραφές και τα λοιπά, κάτι πιο ευέλικτο. Να μην περιοριστούμε δηλαδή όσον αφορά δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Τις άλλες τροπολογίες μπορούμε να τις αποδεχτούμε και είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις ώστε να βρεθεί ένας γρήγορος συμβάσμος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Άλλος. Όχι από ό,τι φαίνεται. Α, ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μεταξύ των συγκητών. Ωραία. Φαίνεται ότι και άλλοι σκιώδεις λείπουν. Ένα πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό έφτασε κάπως καθυστερημένο, αλλά τι να κάνουμε. Μήπως θα θέλατε να πείτε κάτι καταλήγοντας. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το 12-2 την τροπολογία Λάμπερτ. κατά πόσο θα έχουμε δηλαδή ένα κοινό κείμενο ή ε, όχι, δεν ξέρω, αυτό θα μπορούσαμε, αν υπάρχει το κοινό το αποφύγουμε σαν πρόβλημα, αλλά θα το συζητήσουμε βέβαια τους αδέλφους, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. 26 Νοέμβρη θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ. 1η Δεκέμβρη στη ΛΙΤ και θα πάει στην Ολομέλεια του Γενάρη του ερχόμενου Ωραία, ωραία. Καταφωνεί. Έχουμε να κάνουμε τώρα με το θέμα που αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Ο κ. Μπέζες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενθουσιασμός βλέπω. Στην αλλά Αυτό εγώ, αυτό εγώ. Επειδή δεν σα ειδοποίησα σήμερα το πρωί και στο συγγνώμη που έφτασα στο τέλος της μέρας, τι να κάνουμε. Α, για να δω, υπάρχει κανεί που να έχει μείνει και να διαφέρει το θέμα. Δεν βλέπω κανένα. Α, ο κ. Ευτυχώς που έχω και την κούε που με στηρίζει, αλλιώς θα ήμουν θεομόναχος. Και εσά, και εσάς, πρόεδρε, και εσά Πάντω θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να αφήσουμε χρόνο για να συντάξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και δεν είχαμε ιδιαίτερε δυσκολίες εδώ. Συνεργαστήκαμε με τους κοιόδης, περιλάβαμε τα κυριότερα σημεία του κειμένου για να δούμε κατά πόσο είχαμε κάποιες συμφωνίες. Να επιθυμίσω ότι η, η βούληση του Σιγή, βλέπετε το μιλάω στο τρίτο πρόσωπο, είναι το κείμενο αυτό να λάβει σώμα και μορφή πολύ σύντομα και γι' αυτό ακριβώ υπενθυμίζω διαχωρίζουμε τα θέματα που αφορούν την εποπτεία που είναι μέσα στο κείμενο τη Κομισιόν για το οποίο ε, θα πρέπει να εργαστούμε από τα υπόλοιπα θέματα τα οποία αφορούν τι υπόλοιπε τις ε, ε, υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης, αμοιβέ, κρατικό χρέος, δημιουργία ενδεχόμενη οίκου αξιολόγηση ευρωπαϊκού κλπ. Όλα αυτά τα οποία θα είναι ε, θα είναι αντικείμενο της γνωμοδότησης, της έκθεσης μάλλον του Βολτ Κλίμ. Και θα το έχουμε αυτό το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Αυτά που εξετάζω εγώ αφορούν άμεσα βέβαια τα θέματα της εποπτείας που συζήτησε το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του κανονισμού του 2009. Να σας αναφέρω σύντομα τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να λάβουμε θέση. Πρώτο σημείο, διευκρίνηση του όρου χρήσης, της έννοιας χρήσης των συστημάτων εγγύησης όσον αφορά τίτλους που εκδίδονται σε τρίτες χώρες. Κάτι το οποίο ήταν αντικείμενο παρανοήσεων και παρερμηνιών Θα πρέπει να εξετάσουμε επίση το θέμα Τη επικύρωση. τίτλων που εκδίδονται σε χώρε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση και δεν υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρακτικά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε δύο περίοδους. Μία περίοδο κατά τη διάρκεια τη οποία. ο Ευρωπαϊκός Οίκος εξολόγηση θα μπορούσε να επικυρώσει ε, τίτλους οι οποίοι εκδίδονται εκτός Ευρώπης και επικυρώνονται από τους τρεις μεγάλους οίκους εκτός Ευρώπης και μετά δεύτερη περίοδο μέχρι 2011 όπου οι τίτλοι δεν θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο σε περίπτωση που η εξολόγηση φορέα εκτός Ευρώπης ανταποκρινόταν σε συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε λοιπόν τα δύο και θα πρέπει να έχουμε κάποιες ευκρινήσεις. Και αυτά ήταν εξάλλου και ε, αντικείμενο, αυτά τα θέματα αντικείμενο συμβαστικών τροπολογιών. Δομημένα προϊόντα και οι πληροφορίες που παρέχονται για αυτά τα προϊόντα στους οίκους αξιολόγησης και η πρόσβαση στους οίκους αξιολόγησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πληροφόρηση στους οίκους αξιολόγησης ώστε να δίδεται μία άμεση και αυθόρμητη αξιολόγηση. Αυτό μας επιτρέπει βεβαίω να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό και να υπάρχει μία πολυμορφία αξιολόγησης. Αυτό το κείμενο ήταν το κείμενο συζήτησης γιατί είπαν κάποιοι ότι το ίδιο κείμενο το κάνουν και οι Αμερικανοί, δεν είναι πολύ καλό και δεν έχει αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα ότι ρεαλιστικά οι οίκοι αξιολόγηση που δρούν στην Αμερική είναι αυτοί που δρούν και στην Ευρώπη. Θα έλεγα να αφήσουμε αυτό το κείμενο να υπάρχει αυτό της Κομισιόν και να κάνουμε μια αξιολόγηση του κειμένου αυτού πριν από την 1η Ιούλη 2012 και να προβλέψουμε μια ρήτρα αναθεώρηση πριν από τον Ιούλιο του 2014 να δούμε δηλαδή κατά πόσο αυτές οι διατάξεις τήρησαν τους στόχους που τους δόθηκαν όσον αφορά δηλαδή την, τον, την νομοθεσία. Άλλο στοιχείο συζήτησης, δικαιοδοσίες ΕΣΜΑ και κάποιοι είπαν σωστά επ' αυτού ότι δεν έχουμε μόνο τρεις, τρεις οίκους παγκοσμίω, έχουμε και μικρούς οίκους αξιολόγηση στις διάφορες χώρες. Φαίνεται ότι το ΕΣΜΑ δεν έχει πολλούς συνεργάτες ή υπαλλήλου ώστε να κάνει αυτή τη δουλειά το ΕΣΜΑ και να, να χρειάζεται αντίστοιχα ή κατά συνέπεια να κάνουν αυτή τη δουλειά οι, εθνικές, ε, εθνικοί οίκοι Δεν θα πρέπει όμως να εξαρθρώσουμε το έσμα και να αφήσουμε πλήρη αρμοδιότητα στους εθνικούς οίκους αξιολόγησης ανεξαρτήτως της ποιότητάς τους. Αυτό λοιπόν προτείνω και από αυτού υπάρχει ευρεία συμφωνία είναι να έχει δυνατότητα το έσμα να μπορεί να αφήνει συγκεκριμένε αρμοδιότητε στις αρμόδιες αρχές όπως ας πούμε έλεγχος, εποπτεία, επαλήθευση κάποιων στοιχείων κλπ. Και αν επιτρέπετε να πω κάτι παραπάνω, να πω ότι ένας από τους λόγους μπλοκαρίσματος αυτής, τη πρόταση πρότασης είναι ότι οι εθνικές αρχές, δεν με το πει αλλά κάποιοι άλλοι, οι εθνικές αρχές λένε ναι, ναι, εντάξει, πολύ ωραία, ε, εξουσιοδοτείται αυτέ τι αρμοδιότητε, αλλά τι θα μα κοστίσει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα θέμα κατανομή ε, φόρων μεταξύ ΕΣΜΑ και εθνικών αρχών. Και ελπίζω ε, ότι αυτό δεν θα μπλοκάρει τέλο πάντων τι δημόσιε αρχέ. Ένα άλλο θέμα θα πρέπει να ρυθμίσουμε είναι το ποιο θα έχει την αρμοδιότητα για να επιβάλλει κυρώσει στους οίκους αξιολόγησης που διαπράττουν τακτικές παραβάσεις. Νομίζω ότι για νομικούς λόγους ε, συνετά θεώρησε η Κομισιόν ότι αυτή θα έπρεπε, η Κομισιόν δηλαδή θα έπρεπε να επιβάλλει τις κυρώσεις, η λογική λέει θα πρέπει αυτός που ελέγχει να επιβάλλει και κυρώσεις. Ε, σήμερα νομίζω θεωρούμε έτσι σφαιρικά σκεπτόμενοι ότι θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία για επιβολή κυρώσεων και το ΕΣΜΑ. Αυτά λοιπόν σε σχέση με αυτό το θέμα Τώρα, νομίζω ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα συλλογικά σώματα και από τι εθνικέ αρχέ θα πρέπει η μεταφορά αυτή να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Με έναν τρόπο ρεαλιστικό νομίζω ότι η προθεσμία της Κομισιόν 1η 2011 είναι αποδεκτή. Θα μπορούσαμε να πούμε και 1η Γενάρη, αλλά δεν θα ήταν και τόσο ρεαλιστικό να γίνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα στόχο το οποίο θα μπορούσαμε να τηρήσουμε ως προθεσμία. Και βεβαίως στο κείμενο θα πούμε ότι η καταγραφή των αρχών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, η καταγραφή των οίκων αξιολόγησης, θα πρέπει να γίνει όταν, μέχρι να γίνει η μεταφορά του 2011, αυτή η καταγραφή θα πρέπει να είναι ε, σωστή, θα πρέπει να υπάρχει ένα έδος αδειοδότησης και όταν υπάρχει αδειοδότηση θα πρέπει να ξαναγίνει η διοικητική διαδικασία. Θα ήταν λοιπόν καλό το ΕΣΜΑ να κάνει και αυτό ένα έλεγχο όλων των οίκων αξιολόγηση πριν από το 2014 και ούτως ή άλλως ο ρόλος του ΕΣΜΑ με την υποστήριξη των εθνικών αρχών για τον έλεγχο των ελεκτικών αρχών θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο τέλο πάντων βεβαίω ε, ο οίκος αξιολόγησης ε, αξίζει την αδειοδότησή του και την καταγραφή του στο μητρό. Διαφορετικά θα πρέπει να φερείται από το μικρό τη στιγμή που θα τηρεί τις προδιαγραφέ ποιότητα και άλλε προδιαγραφέ που υπάρχουν. Αυτά, Πρόεδρε, σε σχέση με τα σημεία με τα οποία προετοιμάζουμε συμβαστικέ προτάσει. Θα σα τα στείλω όλα αυτά στο τέλο εβδομάδα ή στι αρχέ τη επόμενη για να σκεφτείτε και βεβαίω είμαι ανοιχτό για συζήτηση με του μεν και του δε και προβλέπεται η, ψήφο, η ψηφοφορία στις 22 του Νοέμβρη και Στρασβούρο Δεκέμβρη. Ελπίζω να καταλήξουμε οριστικά τις εργασίες μας ώστε η δικαιοδοσία η υποπτική του ΕΣΜΑ να εφαρμοστεί το ταχύτερο πριν δηλαδή από τη θέση λειτουργία του 2011. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκοζές. Θέλετε εσείς να πείτε κάτι, παρακαλώ. Τι να πω τώρα εγώ. Να πιούμε ένα καφεδάκι και να τα πούμε μετά. Ε, λοιπόν, όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα τώρα. Εντάξει. Θα έλεγα, είχαμε συμφωνήσει ούτω ή άλλω εν μέρη και όταν θα έχουμε τι συμβιβαστικέ τροπολογίε μπορούμε να παραμείνουμε σε επαφή και να τα συζητήσουμε. Κατά τα άλλα μπορώ να εγκρίνω αυτή την αρχή την οποία εσύ παρουσίασες. Okay, so I understand you know... Εντάξει. Λοιπόν, θα διανεμηθούν αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες σύντομα, έτσι. Fine. Well, I just... Πολύ καλά. Επαναλαμβάνω τις ημερομηνίες που ανέφερε ο κύριος Γκορζές 22 Νοεμβρίου ψήφιση στην Επιτροπή και μετά θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο προ συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτά για σήμερα. Επόμενη συνεδρίαση. Η ημερομηνία επόμενη συνεδρίασης, 22 Νοεμβρίου. Σημειώστε το παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Γεια.